Να ξαναρχίσουμε τη συνεδρίασή μα. Η ακρόαση σήμερα το απόγευμα έχει να κάνει με τι τρίτε χώρε για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Στο πλαίσιο του πρώτου κλάστερ, Έχουμε τον τίτλο «Η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων υπό το φως του οργανωμένου κλίματος» και θα ακούσουμε την κυρία Μυρία Βασιλιάδου, η οποία είναι συντονίστρια κατά της εμπορίας ανθρώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν ε, να δώσω το λόγο στην κυρία Βασιλιάδου, ε, έπρεπε να κάνω μια ανακοίνωση. Σε λίγα λεπτά θα εγκαταλείψω την Προεδρία, γιατί πρέπει να μεταβώ στην Ιταλία αύριο το πρωί. Θα είμαι στη δικαστική αίθουσα, θα με εξετάσει ένας δικαστής, γιατί πριν δύο χρόνια, νομίζω ότι γνωρίζετε πολύ τον ε, Τωρίνα, ο οποίος είναι επικεφαλής ε, της Ιταλικής Μαφίας, πριν ε, δύο χρόνια με απείλησε με θάνατο, έτσι αύριο θα καταθέσω στο δικαστήριο και θα πρέπει να εγκαταλείψω την αίθουσα για να μεταβώ στο αεροδρόμιο, να φτάσω στο Μιλάνο και έτσι αύριο το πρωί να παρευρεθώ στο δικαστήριο. Σας ζητώ λοιπόν συγγνώμη κυρία Βασιλιάδου, δυστυχώς ε, με καλεί το καθήκον. Φυσικά ως πολιτική αγωγή θα καταθέσω. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση. Έχετε 15 λεπτά για την παρουσίασή σας και στη συνέχεια θα περάσουμε στη συζήτηση με τους συναδέλφους. Παρακαλώ. Thank you. Thank you very much for, for inviting me. Ευχαριστώ που με καλέσατε σήμερα. Έχω παρευρεθεί σε αρκετές ακροάσεις στο Κοινοβούλιο την προηγούμενη διετία μετά το διορισμό μου. Πρώτη φορά έρχομαι όμως στην Επιτροπή σας. Ευχαριστώ για την ε, πρόσκληση, ευχαριστώ ιδιαίτερα την κυρία Αλφάνου. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπαιξε ζωτικό ρόλο για το, την διαμόρφωση της απάντησης της Ένωσης στην εμπορία ανθρώπων όπου υπάρχει ανάληψη δέσμευσης νομίζω, όπου υπάρχει πολιτική υποστήριξη, γίνονται πράγματα και έχουμε καλύτερη και συνολικότερη απάντηση, η οποία σε τελευταία ανάλυση κάνει διαφορά στις ζωές των θυμάτων. Να ευχαριστήσω την κυρία Αγιάλα για το θεματικό έγγραφο. Είχαμε επικοδομητική συνεργασία, την ευχαριστώ γι' αυτό και εκτιμώ τη συνεργασία. Και για να αρχίσουμε από τα βασικά, θα ήθελα να θυμηθούμε όλοι σήμερα ότι όταν μιλάμε για εμπορία ανθρώπων θα μπορούσε να είναι κάτι που γίνεται και στη διπλανή πόρτα. Μπορεί να γίνει στη γειτονιά μας και πρόκειται για τη σύγχρονη δουλεία. Είναι σοβαρή ε, παραβίαση ανθρωπίνων ελευθεριών, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και είναι σοβαρή μορφή οργανωμένου εγκλήματος. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας πριν από έξι μήνες μόλις έδωσε στοιχεία για την περίοδο 2002-2011 και μιλάει για μέχρι και 21 εκατομμύρια θύματα ε, αναγκαστικής εργασίας σε όλο τον κόσμο και 5,5 εκατομμύρια από αυτά υπολογίζουν ότι είναι παιδιά και περίπου 880.000 είναι στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχίσαμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα, για πρώτη φορά γίνεται αυτό, για τη συλλογή δεδομένων σε επίπεδο ένωσης. Εσείς ε, θα γνωρίζετε στην Επιτροπή σας πόσο δύσκολη είναι η συλλογή στοιχείων για τέτοιες κρυφές μορφές εγκλημάτων και ότι δεν είναι πολύ αξιόπιστα πάντα τα στοιχεία αυτά, αλλά πάντως υπάρχει η γενικότερη κατεύθυνση να φροντίσουμε να βρούμε πιο αξιόπιστα στοιχεία που θα συλλέγονται με καλύτερο τρόπο σε όλη την Ευρώπη. Αυτό που είδαμε λοιπόν και η έκθεση θα δημοσιευτεί τους επόμενους δύο μήνες ελπίζω, είναι ότι έχουμε 76% των θυμάτων που είναι θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, μιλάω για το 2010, τα υπόλοιπα είναι θύματα που, αναγκαστικής εργασίας, ε, αναγκαστικής επαιτίας και πετία στο σπίτι η ε, σύγχρονη δουλεία στα σπίτια. Σύγχρονα νέα κορίτσια είναι το 79% και 21% οι άνδρες. 3% είναι ε, αγόρια και 12% κορίτσια. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι η εσωτερική ε, διακίνηση αυξάνεται ε, ξέρω τα σημερινά μας θέματα, αλλά ας θυμηθούμε ότι σε μεγάλο βαθμό η εσωτερική διακίνηση υπάρχει. Βλέπουμε λοιπόν ότι και μέσα στο έδαφος της Ένωσης διακινούνται παράνομα. Και τα περισσότερα θύματα από τρίτες χώρες έρχονται από την Ιγυρία και την Κίνα, από ό,τι φαίνεται. Και αυτό συνάδει και με τα τελευταία ε, δεδομένα ε, τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την ποιότητά τους, τον αριθμό τους και την κατηγορία δεδομένων έχει βελτιωθεί πολύ από το 2008 όπου άρχισε η πρώτη συλλογή δεδομένων μέχρι το 2010. Οπότε νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Και επίσης ε, έχουμε και μια οδηγία για την εμπορία ανθρώπων που προβλέπει ότι οι αρμόδιοι εθνικοί μηχανισμοί πρέπει να συλλέγουν αυτά τα δεδομένα υποχρεωτικά. Η εμπορία ανθρώπων είναι σύνθετο φαινόμενο υπερεθνικό. Μιλάμε για ανθρώπους που τους πουλούν στις οικοδομές, στη γεωργία, στην κλωστοϊφαντουργία, ε, στα ε, οσικιακή βοηθή. Υπάρχει μακρύς κατάλογος. Ε, πολλές φορές αφαιρούνται όργανα, γίνονται παράνομες υιοθεσίες, ε, αναγκάζονται να συμμετέχουν σε εγκληματικές δραστηριότητες κλπ. Και ξέρουμε ότι και τα κράτη-μέλη συμφωνούν ότι είναι μια μορφή εγκλήματος όπου δεν μπορούν να δράσουν μόνο τους τα κράτη-μέλη. Χρειάζεται νοσιακή δράση. Και αυτό αντικατοπτρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην οδηγία, στην φιλοδοξία που έχει η οδηγία που θεσπίσαμε. Έτσι λοιπόν θα σας δώσω κάποια ε, θέματα για τους τομείς δραστηριοτήτων της Ένωσης. Ό,τι αφορά το νομοθετικό το επίπεδο, έχουμε την οδηγία από το 2011 η οποία προλαμβάνει και καταπολεμεί την διακίνηση και προστατεύει τα θύματα. Ε, είναι ποινική νομοθεσία, θα λέγαμε, στα πλαίσια της συνθήκης Λισαβόνας. Πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι το πρώτο αυτό. Τι κάνει, αναρμονίζει τον ορισμό του, του, εγκλήματος και τις ποινές και έχει στεναρές διατάξεις για την δίωξη των διακινητών, επικεντρώνεται δε και στην προστασία, υποστήριξη, αρρωγή των θυμάτων. Αυτά τώρα για την νομοθεσία. Για την πολιτική θα επανέλθω και αργότερα. Τώρα όμως έχουμε τη στρατηγική της Ένωσης για την εξάλληψη της διακίνησης ανθρώπων και την εμπορία τους για την περίοδο 2012-2016 που περιλαμβάνει 40 συγκεκριμένες πολιτικές δράσεις μαζί με την οδηγία, παράλληλα με την οδηγία, έχουμε και συμπεράσματα του Συμβουλίου που εγκρίθηκαν πέρσι τον Οκτώβριο και που δίνουν στεναρό μήνυμα πολιτικής στήριξης και καλούν τα κράτη-μέλη μεταξύ άλλων να διασφαλίσουν την έγκαιρη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο της οδηγίας. Και έχουμε και χρηματοδότηση και εδώ και όλα, αυτά τα χρόνια η Κομισιόν στήριξε πολλά προγράμματα, πολύ άριθμα για την εμπορία ανθρώπων. Πέρσι που κάναμε ε, συλλογή όλων των προγραμμάτων που χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχουν 11 γενικές ε, διευθύνσεις που χρηματοδοτούν ε, τέτοια προγράμματα για την εμπορία ανθρώπων και υπάρχουν αυτά σε ένα ειδικό website, υπάρχουν όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από το 2003-2004 και μετά από τις διάφορες υπηρεσίες. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα στο DG Εσωτερικές Υποθέσεις για τα, την εμπορία οργάνων και άλλα, και, άλλους, και άλλα μέσα όπως διαχείριση μεταναστευτικών ορών, ε, το πρόγραμμα Δάφνη για τη βία των γυναικών, μετανάστευση άσυλο κλπ. Αυτά για να σας δείξω ότι και πάλι η εμπορία ανθρώπων είναι, ένα, ε, είναι μια μορφή οργανωμένου εγκλήματος, αλλά έχει και άλλες διαστάσεις που τις ε, μελετούν όλες αυτές οι χρηματοδοτικές δυνατότητες. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν με όλα αυτά τα προγράμματα, τα, τα έργα, γιατί είναι πολλά, αν δείτε και την ιστοσελίδα, το 2014 πρόκειται να κάνουμε μια ε, συνολική ανασκόπηση όλων αυτών που χρηματοδοτήσαμε για να δούμε ε, από πού προέρχεται και πού οδηγεί μια πολιτική και να έχουμε καλύτερη ε, αντιστήχηση στις χρηματοδοτήσεις σε σχέση με τις πολιτικές προτεραιότητες. Σε αυτή την οδηγία λοιπόν για τη διακίνηση προς ανθρώπων, την εμπορία ανθρώπων, υπάρχει ένα άρθρο για το, τη θέση που κατέχω και αυτό είναι κομμάτι του προγράμματος Στοκχόλμης, αρχικά δηλαδή από εκεί προήλθε από το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Θα εξηγήσω σε δύο λεπτά τη δική μου την εντολή. Επίσης θέλω να σας πω ότι μιλάμε για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και αυτό είναι κάτι που απασχολεί και αυτή και άλλες επιτροπές. Προσπαθούμε να μην μιλάμε για καταπολέμηση, αλλά για την ε, ενασχόληση της ε, εμπορίας, γιατί θέλουμε να συμπεριλάβουμε εκτός από τη δίωξη και την πρόληψη. Αυτό που κάναμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν για να έχουμε μια πιο συνεκτική προσέγγιση είναι να συμπεριλάβουμε και ζητήσαμε από 17 ε, υπηρεσίε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνέρχονται τώρα διπηρεσιακά από την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επιχειρήσει, τη δικαιοσύνη, την υγεία, την εκπαίδευση και πολλές άλλες διευθύνσεις να συμβάλλουν σε αυτό το πλαίσιο πολιτικής και συμβάλαμε με πάνω από 13 εσωτερικές διαβουλεύσεις για να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει συνοχή στους επιμέρους τομείς πολιτικής μας. Ε, αυτή η στρατηγική της Ένωσης επικεντρώνεται γύρω από πέντε βασικούς τομείς ε, να εντοπίσουμε, να προστατεύσουμε τα θύματα, να προλάβουμε την εμπορία, μείωση των απαιτήσεων, αυτό αναφέρεται και στο έγγραφο της κυρίας Αγιάλα, ε, βελτιωμένη δίωξη, καλύτερο συντονισμό και συνεργασία και καλύτερη αντίδραση στο έγκλημα αυτό. Σε σχέση με τις τρίτες χώρες, τα κράτη-μέλη ενέκριναν τώρα τη δεύτερη έκθεση ε, εφαρμογή για την εξωτερική δράση της Ένωσης στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων. Αυτό ήταν πολιτικά ευαίσθητο θέμα. Καταρτήσαμε έτσι ε, τρίτες χώρες ε, που δυσανάλογα πλήττονται από την εμπορία προσώπων και εκεί θα επικεντρώσουμε την εξωτερική μας δράση. Αυτό λοιπόν ήταν ε, προτεραιότητα εδώ και χρόνια, γιατί θέλουμε μια πιο στρατηγική προσέγγιση. Επί Σουηδικής Προεδρίας το Συμβούλιο ενέκρινε αυτό το έγγραφο με προσανατολισμό τη δράση και εδώ έχουμε τα αποτελέσματα της δεύτερης ε, έκθεσης πεπραγμένων. Έχουμε κατάλογο 10 χωρών προτεραιότητας και χώρες με τις οποίες θα συνεργαστεί περισσότερο η Ένωση. Η στρατηγική της Ένωσης ε, κυρίως ε, βασίζεται στα θύματα και επειδή επικεντρώνεται στα θύματα προετοιμάσαμε τώρα και θα δημοσιευτεί πολύ σύντομα ε, σαφείς πληροφορίες ε, φιλικές προς το χρήστη για τα δικαιώματα στα πλαίσια του ενωσιακού δικαίου των θυμάτων. Σύντομα θα δημοσιευτεί και θα μεταφραστεί στο Εθνικό Δίκαιο το 2014, στο εσωτερικό δίκαιο κάθε χώρας. Επίσης θέλουμε και πλατφόρμα ε, υπηρεσιών για τα θύματα που λειτουργούν όπως πρέπει στα κράτη-μέλη και στην Ένωση. Αυτή η πλατφόρμα θα αρχίσει να λειτουργεί Μάιο-Ιούνιο φέτος και θέλουμε να προσέξουμε πολύ και το θέμα της ζήτησης των υπηρεσιών από τα θύματα της ε, εμπορίας. Υπάρχει τώρα για 2,5 εκατομμύρια ευρώ ένα αίτημα από την Γενική Διεύθυνση Έρευνας για να ασχοληθεί με το θέμα και ελπίζουμε ότι θα συμβάλλει στην πολιτική για το 2016. Σε αυτό το θέμα θα επανέλθω σε ένα λεπτό. Επίσης θα αρχίσουμε και ε, μια συμμαχία επιχειρήσεων το 2014 κατά της εμπορίας προσώπων για να δουλέψουμε με τον ιδιωτικό τομέα. Μίλησε για την κοινωνία των πολιτών, την επιχειρηματική κοινότητα, τον ιδιωτικό τομέα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διεθνείς Οργανώσει, συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Επίσης δουλεύουμε και με φορείς δικαιοσύνη και εσωτερικών υποθέσεων ε, ότι η μέρα που διοργανώσαμε ε, στις 18 Οκτωβρίου, τη μέρα κατά το σωματεμπορίας, 18 ε, φορείς συναντήθηκαν στην Βαρσοβία και υπέγραψαν κοινέ δηλώσει, υπέγραψαν οι, διευθυντές, οι ε, για τα θέματα αυτά και τι θα κάνουν. Και στη στρατηγική είπαμε ότι πρέπει τώρα να υλοποιήσουμε αυτέ τι δεσμεύσει. το κάνουμε, έχουμε σημεία επαφή, συνδέσμους που συνέρχονται κάθε δύο-τρει μήνε για να συζητήσουν τι δράσει του. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο το εγχείρημα, διότι ε, υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη συνοχή, γιατί τώρα υπάρχουν πολλές παράλληλες εργασίες και δεν συλλέγονται πολλές πληροφορίες, αλλά εμείς ε, προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε. Για να επικεντρωθώ λίγο περισσότερο στα θέματα που σας ενδιαφέρουν εσάς ως Επιτροπή περισσότερο. Η πιο ανησυχητική τάση στην εμπορία προσώπων είναι ο χαμηλός αριθμός των διώξεων. Πολύ χαμηλές, ανησυχητικά χαμηλός αριθμός. Η τρίτη προτεραιότητα της στρατηγικής προβλέπει αυξημένη δίωξη των διακινητών είναι πολύ προσοδοφόρο σε εγκληματική δραστηριότητα, 32 δις δολάρια, 25 ε, δις ευρώ είναι τα κέρδη για τους διακινητές ετησίως και Πρέπει βέβαια να τους αφαιρέσουμε τα οικονομικά κίνητρα και να χτυπήσουμε τα δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος που διευκολύνουν όλα αυτά. Και γι' αυτό στη στρατηγική μας λέμε ότι χρειάζονται οικονομικές έρευνες. Για, όχι μόνο γιατί έτσι θα έχουμε και αποδείξεις στο δικαστήριο για την ε, αποτελεσματική δίωξη, αλλά θα μετριάσουμε και το οικονομικό όφελος και θα βελτιώσουμε τις έρευνες ε, που θα μας δίνουν πληροφορίες για τα εγκληματικά δίκτυα. Αυτή η διεθνική ε, διάσταση του εγκλήματος πρέπει να μας απασχολήσει. Και μπορούμε στις μονάδες ε, πληροφόρησης της Ένωσης μπορούμε να βρούμε ε, βοήθεια και συνεργασία. Μπορεί να υπάρχει επίσης αξία ε, από την εναρμόνιση του αδικήματος, του ξεπλήματος χρήματος σε ενωσιακό επίπεδο. Και συναφές ε, πεδίο είναι η προτινόμενη οδηγία για το πάγωμα και τη δίμευση των, προσ... εσόδων εγκλήματος που θα διευκολύνουν τις αρχές των κρατών μελών να δημεύουν και να παίρνουν πίσω τα έσοδα από το διασυνοριακό σοβαρό έγκλημα. Ένα άλλο φαινόμενο που το οποίο συζητείται πάρα πολύ είναι η διαφθορά. Τώρα ετοιμάζομαι μια έκθεση κατά της διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ε, υποβάλλεται κάθε δύο χρόνια, θα εκδίδεται και για πρώτη φορά αυτό θα γίνει φέτος. Η αξιολόγηση της απειλής ε, ε, και η σχετική έκθεση αναφέρει ότι στην εμπορία ανθρώπων ε, οι πιο απειλητικές ομάδες είναι αυτές που μπορούν να ελέγξουν όλη τη διαδικασία της διακίνησης συμπεριλαμβανομένου του ξεπλήματος χρήματος και υψηλού επίπεδου διαφθορά. Τέλος, Έχουμε το impact που είναι ε, η αναφορά για το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η προτεραιότητα S αφορά ακριβώς την εμπορία ανθρώπων. Και αυτό που είναι ενδιαφέρον και πολλά υποσχόμενο είναι ότι η Europol επιβεβαίωσε ότι ο αριθμός των εισφορών των κρατών μελών έχει διπλασιαστεί σε σύγκριση με την ανάλογη περίοδο πέρσι. Τώρα δηλαδή έχουμε ροές πληροφοριών στο 100%. Εντυπωσιακέ πληροφορίες έχουν δοθεί και ανταλλαγή μεταξύ κρατών μελών και Europol και πολλά άλλα θετικά. Οπότε έχουμε τα εργαλεία, έχουμε τις πολιτικές στη διάθεσή μας, έχουμε και χρηματοδοτικά μέσα. Ελπίζω ότι θα έχουμε και πολιτική στήριξη για να δώσουμε συνέχεια σε όλα αυτά τα θέματα. Προσβλέπω στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βεβαίως και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα αναρωτιέστε πόσοι εδώ εκτελούν χρέη Προέδρου. Δυστυχώς, όπως ακούσατε, πρέπει η Πρόεδρος να στρέψει σήμερα στην Ιταλία. Ζητώ συγγνώμη, λοιπόν, γι' αυτό. Έχω εδώ την κυρία Αγιάλα, καταρχήν. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Βασιλιάδου. Επίσης, ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, καλή συνεργασία που είχαμε για να συντάξουμε την έκθεση για την εμπορία ανθρώπων στο πλαίσιο αυτή της Επιτροπής. Ακριβώς ε, τη στιγμή που άρχιζε ε, να τίθεται σε λειτουργία η οδηγία. Νομίζω ότι φέτος, ε, το Μάρτιο, θα πρέπει να δούμε τι έχει γίνει με τη μεταφορά στο ιστορικό δίκαιο και με ποιο τρόπο μπορεί να λειτουργήσει. Και μάλιστα τη στιγμή που ξεκινούσε και η στρατηγική 2012-2016 για τις νέες δράσεις ε, που πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή για να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο. Επίσης, εσείς μας δηλώσατε δύο πτυχές, ε, η εμπορία ανθρώπων καταρχήν για σεξουαλική εκμετάλλευση και δεύτερον ε, το θέμα της ε, εργασιακής εκμετάλλευσης. Έχουμε λοιπόν δύο όψεις αυτού του φαινομένου, τρομακτικές όψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αφού Αναθεωρήσαμε όλα τα κύματα και πραγματικά μου ανοίξατε τα μάτια και επί όλων των εκθέσεων της Ευρωπόλ που ήταν ιδιαίτερα αποφασιστικές και τις μαρτυρίες ε, από τους οργανισμούς. Η εντύπωση που έχουμε είναι ότι δεν μειώνεται το φαινόμενο, το αντίθετο μάλιστα αυξάνεται. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η τάση παρόλο που έχουμε περισσότερα ευρωπαϊκά μέσα και περισσότερες δράσεις, δυστυχώς φαίνεται ότι δεν μπορούμε να περιορίσουμε τη ζήτηση. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, δηλαδή τι δράσεις θα μπορούσαμε να λάβουμε για να μειώσουμε τη ζήτηση εσείς. Αναφερθήκατε και σε ένα λεπτό ε, θέμα, δηλαδή να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα και με τρίτες χώρες, γιατί ο σεξουαλικός τουρισμός ε, είναι πραγματικά μια σταγόνα στον ωκεανό. Τη εμπορία ε, ανθρώπων και για σεξουαλική εκμετάλλευση και για εργασική εκμετάλλευση. Εγώ λοιπόν ήθελα να σας ρωτήσω αν στη συνεργασία σας με τρίτες χώρες για τον περιορισμό του φαινομένου λαμβάνονται υπόψη και οι κυρώσεις, τι είδους κυρώσεις θα υπάρξουν. Δηλαδή θα πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις, ποινές στους ανθρώπους αυτούς και αυτό θα πρέπει να το λαβούμε υπόψη και όταν υπογράφουμε συμφωνίες με τρίτες χώρες. Δηλαδή, εμείς ε, να μην συνάπτουμε συμφωνίες που επιδεινώνουν, οικονομικές μόνο συμφωνίες που επιδεινώνουν ε, το φαινόμενο αυτό και επίσης να δούμε και τι θα κάνουμε με το θέμα της ζήτησης. Έχουμε μια τρομερή κατάσταση, πολύ μεγάλη διακίνηση και εμπορία τέτοιων ανθρώπων και εμείς που έχουμε αγωνιστεί για ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και για την εξάλληψη της εκμετάλλευσης, δυστυχώς βλέπουμε να υπάρχει μία ζήτηση για σεξουαλική εκμετάλλευση. Όμως και σε κατάσταση κρίσης, σε καιρούς κρίσης. Επίσης, βλέπουμε να υπάρχει ζήτηση για ε, σκλάβους. Ε, ε, δηλαδή προσπαθούμε να τους νομοποιήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, όμως υπάρχουν και κάποιες τρομακτικές πτυχές σε όλο αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, όταν μιλάμε για αξιοπρεπή εργασία και για ποιότητα ζωή, σε πολλέ φορές βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν αξιοπρεπεί συνθήκε στην εργασία. Για μιλάμε για εργασιακού σκλάβου. Έτσι λοιπόν, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω αυτά τα δύο. Ποιες κυρώσεις βλέπετε στα πλαίσια της Συνάψης Συμφωνίας και Συνεργασίας με τρίτες χώρες και σε σχέση με τις καταδίκες ε, όσων προβαίνουν σε νομοποίηση παρανόμων εσόδων και τι θα κάνουμε και για τη μείωση της ζήτηση. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να θέσουμε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο και να απαιτήσουμε να υπάρχουν κυρώσεις ε, και να υπάρχουν και καταδίκες δηλαδή να αρχίσουμε να εργαζόμαστε για να εφαρμόσουμε τον νόμο πλήρως. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νιτοντάν. Thank you. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα. Η, την ποιότητα της Επιτροπής μας πρέπει να προσέχετε έτσι, όχι την ποσότητα εδώ. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Εγώ έχω πέντε ερωτήσεις. Μία είναι Πώς συνεργάζονται τα κράτη-μέλη μαζί σας, συνεργάζονται με τον ίδιο τρόπο όλα ή όχι. Δεύτερον, η συνεργασία η διασυνοριακή μεταξύ των χωρών μελών λειτουργεί καλά ή υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή υπάρχουν καθυστερήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Τρίτον, είπατε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι θύματα παράνομης διακίνησης έρχονται από την Ιγυρία, την Κίνα Εντάξει, ξέρω ότι στη θεωρία υπάρχει η ελεύθερη διακίνηση, αλλά τι σημαίνει αυτό. Τέταρτον, κάτι πολύ ενδιαφέρον που είπατε, ότι οι διώξει είναι πολύ χαμηλέ. Ο αριθμό των διώξεων. Γιατί δυσκολεύεστε να έχετε αποδείξει, ποιο είναι το πρόβλημα εκεί. Και πέμπτον, όπως ξέρετε, η Επιτροπή μας θα καταλήξει σε μία έκθεση με συστάσεις για το πώς θα μπορέσει καλύτερα να καταπολεμήσει η Ευρώπη τα φαινόμενα αυτά που συζητάμε. Λοιπόν, τι συστάσεις θα είχατε να κάνετε στην Επιτροπή μας για να συμπεριλάβει στην έκθεσή της, ότι δηλαδή προτείνεται να γίνει αυτό, εκείνο, το άλλο, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ε, κυρία Ευχαριστώ πολύ. Ήδη αναφέρθηκε το θέμα της ισότητας μεταξύ αντρών και γυναικών. Προφανώς πρόκειτο για την παράνομη διακίνηση με στόχο την σεξουαλική εκμετάλλευση των γυναικών. Ε, προφανώς εκεί τα θύματα είναι οι γυναίκες. Εγώ θέλω όμως να αναφερθώ και σε μια άλλη διάσταση της ισότητας στα πλαίσια και της δια, παράνομης διακίνησης για σεξουαλική εκμετάλλευση αλλά και για ε, εργασιακή εκμετάλλευση. Δεν υπάρχει η ίδια κατάσταση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως μεταξύ τους. Τα περισσότερα θύματα έρχονται από την Ανατολική Ευρώπη ή και από την Νότια. Θα έλεγα είναι δεύτερης τάξης ε, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εκεί μεταφέρονται στις παλιές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί όπου έχουμε τις πιο πλούσιες ε, παραδοσιακές κοινωνίες. Δεν έχω δει ποτέ να γίνεται παράνομη διακίνηση μιας Ολλανδέζας, ας πούμε, που να την παίρνουν από την Ολλανδία και να την πηγαίνουν παράνομα στη Βουλγαρία ή στη Ρουμανία για να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά. Το αντίθετο συμβαίνει. Ούτε βέβαια έχω δει κανέναν Γερμανό άντρα να ζει κάτω από συνθήκες δουλείες στην Ουγγαρία ή στην Ρουμανία. Τι νούμερα έχετε για αυτές τις περιπτώσεις και γιατί υπάρχει πάντα σιωπή σε αυτήν την σημαντική διάσταση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων. Τι στοιχεία έχουμε, ποιες είναι οι αναλογίες. Και ποιοι είναι οι λόγοι και οι αιτίες για την παράνομη αυτή διακίνηση που έχει σαν στόχο την εκμετάλλευση των ανθρώπων, είτε τη σεξουαλική, είτε ε, τους βάζουν να δουλεύουν. Δεν άκουσα όμως αυτό που περίμενα να ακούσω. Δηλαδή όταν μιλάμε για την παράνομη διακίνηση ε, των γυναικών με στόχο την ε, εκπόρνευσή τους, την πορνεία, ίσως πρέπει να δούμε και την ζήτηση που υπάρχει για την πορνεία. Αν δεν υπάρχει ζήτηση, δεν θα υπήρχε. Αν απαγορευτεί δηλαδή, δεν θα υπάρχει. Η θα έπρεπε να υπάρχει και δίωξη των πελατών. αυτόν δηλαδή που τη ζητούν την πορνεία. Άρα λοιπόν την ζήτηση, όταν αναφερθήκατε στη ζήτηση εννοούσατε αυτή την ζήτηση, τη ζήτηση που υπάρχει για την πορνεία και την σεξουαλική εκμετάλλευση των γυναικών. Τι ισχύει σήμερα στην Ευρώπη επίσης για την πορνεία που γίνεται εντό αγωγικών εθελοντικά σε σχέση με αυτήν που δεν γίνεται εθελοντικά, και εγώ δεν πιστεύω και πολύ σε αυτή τη διάκριση. Και ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σχέση της πορνείας με την παράνομη διακίνηση. Ο κύριος Καρόνα, έχω μία απλή ερώτηση και εν μέρη σχετίζεται με όσα ακούστηκαν από την τελευταία ομιλήτρια. Εγώ θα ήθελα να καταλάβω καλύτερα τις διαστάσεις του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων και πιο συγκεκριμένα στην Ευρώπη. Εγώ νομίζω αναφερθήκατε σε 5 εκατομμύρια ανήλικους και σε 580.000 στην Ευρώπη. Θα ήθελα να ξέρω τα νούμερα του φαινομένου της εμπορίας και δεύτερον οι εγκληματικές οργανώσεις που εμπλέκονται σε αυτή την εμπορία. Δηλαδή, ε, από ποιες χώρες συνήθως προέρχονται, δηλαδή ε, είναι ε, άνθρωποι Ευρωπαίοι πήκοοι και αν ναι, σε, ποια χώρες; σε ποιες χώρες βλέπουμε το φαινόμενο, κύριε Μακεντάι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχα κάποιες ερωτήσεις. Δηλαδή, καταρχήν θέλω να πηχήσω αυτό που ρώτησε ο κύριος Νιούτον Ντάν. Γιατί έχουμε τόσο χαμηλό αριθμό διώξεων. Μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχουν διάφοροι λόγοι, αλλά θα ήθελα να ακούσω αν εσείς κατανοείτε καλύτερα το λόγο. Φαίνεται πολύ ενθαρρυντικό το ότι έχουμε 100% αύξηση στις ε, ροές πληροφοριών που έρχονται στη Europol. Και νομίζω η Europol ε, κάνει μια ιδιαίτερα αξιόλογη δουλειά και χαίρομαι ιδιαίτερος. Αναρωτιέμαι αν αυτή η 100% αύξηση από πέρσι οφείλεται σε μεγαλύτερη συνεργασία ή επειδή έχουμε μεγαλύτερη εμπορία υπήρξε και τέτοια αύξηση. Γιατί έχουμε λοιπόν την αύξηση αυτή. Τρίτον, σε άλλες τοποθεσίες ε, είδαμε το θέμα της εμπορίας παιδιών, αν υπάρχει εμπορία παιδιών και πώς ε, μπορεί να γνωρίζει κάποιος ότι υπάρχει εμπορία παιδιών. Ε, εσείς μιλάτε συγκεκριμένα για εμπορία ανθρώπων, όμω όμως μπορείτε να μας μιλήσετε για τα παιδιά πιο συγκεκριμένα και αν προέρχονται από τρίτες χώρες και ναι, από ποιες χώρες. Well, thank you very Ευχαριστώ πολύ για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και όλα αυτά τα ενδιαφέροντα σημεία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορείτε να απαντήσετε. Μπορείτε ίσως ε, να συνοψίσετε ταυτόχρονα και την παρουσίασή σας με τις απαντήσεις που θα δώσετε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω και ελπίζω να τα καλύψω όλα. Να ξεκινήσω με τις τρίτες χώρες. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό. Και λαμβάνοντας υπόψη και το θέμα της σημερινής συνεδρίασης ευρύτερα. Υπάρχουν ε, τα Action Oriented Papers, τα έγγραφα προσανατολισμού δράσης. Αυτά αναπτύχθηκαν το 2009 από τη Σουηδική Προεδρία. Τώρα έχουμε τη δεύτερη έκθεση εφαρμογή που διατήθηκε το Δεκέμβριο του 2012. Τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο τι έκαναν κατέρτισαν ένα κατάλογο χωρών προτεραιότητας. Έχουμε εκεί 10 χώρες, αλλά έχουμε και ένα κατάλογο περιφερειών και κάποιου εταίρου με του οποίου θα θέλαμε να συνεργαστούμε στον τομέα τη εμπορία ανθρώπων. Πώ ε, καταρτήσαμε αυτόν τον κατάλογο, Προέκυψε ω αποτέλεσμα των δεδομένων που είχαμε ε, της δικής μας πιλωτικής ε, συλλογής δεδομένων φέτος ως αποτέλεσμα εκθέσεων από τη Europol, τη Frontex, από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, από το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας και από το UNODC. Έτσι λοιπόν, ε, αυτά τα δεδομένα μας οδήγησαν να πιστεύουμε ότι ιδίω σε αυτές οι δέκα πρώτες χώρες είναι χώρες όπου θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να επικεντρωθεί. Και αυτό τώρα συζητείτε με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση για να δούμε πώ η Κομισιόν μπορεί να συνεισφέρει σε αυτό και πώ μπορούμε να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη για να διασφαλίσουμε πιο εστιασμένη χρηματοδότηση ή άλλε δραστηριότητε για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Για τα δεδομένα. Με ρωτήσατε τι γίνεται με τα παιδιά συγκεκριμένα από τα προκαταρκτικά δεδομένα και πρέπει να πω, όσο είπα στην αρχή, ότι τα δεδομένα είναι ενδεικτικά. Αυτό μας είπαν τα κράτη-μέλη. Η ποιότητα των δεδομένων έχει βελτιωθεί από το 2008 στο 2010, αλλά σε τέτοια ζητήματα θα έλεγα ότι βλέπουμε την κορφή του παγόβουνου. Έχουμε περίπου 15% παιδιά, 12% κορίτσια και 3% γόρια που είναι θύματα εμπορίας και δίνουμε πολύ μεγάλη προσοχή στην Κομισιόν. Θα σας δώσω μία ένδειξη. Θα έλεγα ότι το ίμιση της χρηματοδότησής μας, κυρίως στην δέλτα ιστορικών υποθέσεων, ε, προορίζεται για την αντιμετώπιση της εμπορίας παιδιών. Εργαζόμαστε στενά με την Κομισιόν και τους συναδέλφους ε, στην κατεύθυνση αυτή. Ε, έχουμε μία μελέτη προς ολοκλήρωση από το ICMPD που αφορά την αξιναγκαστική επαιτία. Έχουμε παιδιά. Δεν μπορώ να σας δώσω τώρα νούμερα. Θα δημοσιευτεί όμως ε, η έκθεση αυτή του επόμενους ε, δύο μήνες. Θα έχετε και συγκεκριμένα νούμερα, συγκεκριμένους αριθμούς για τον παιδιά και από πού προέρχονται συνήθως. Ε, κάποια θύματα παιδιά είναι και υπηκοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι αυτό σχετίζεται περισσότερο ότι είναι αντικείμενο εμπορία για να ταωθούν στην εξαναγκαστική επαιτία. Τώρα ολοκληρώνεται αυτό το έγγραφο του SMPD, όπω σα είπα. Τώρα, δεν μπορώ να σα δώσω συγκεκριμένου αριθμού, ε, μακάρι να μπορούσα, αλλά δυστυχώ δεν μπορώ. Και νομίζω ότι γνωρίζετε, ειδικά σε αυτή την Επιτροπή, πόσο δύσκολο είναι να έχουμε αριθμητικά στοιχεία όταν μιλάμε για δραστηριότητες που, είναι, ε, που αφορούν κυρίως το οργανωμένο έγκλημα. Επικεντρωνόμαστε βέβαια σε αυτό, χρηματοδοτούμε αρκετά σχέδια και ε, συνεργαζόμαστε με τους εθνικούς συγητές και τους αντίστοιχους μηχανισμούς στα κράτη-μέλη για να δούμε πώς μπορούμε να συλλέξουμε καλύτερα τα δεδομένα. Ελπίζουμε ότι στο επόμενο εγχείρημα θα επαναληφθεί σε δύο χρόνια αυτό το πιλωτικό project και θα βάλουμε τα δυνατά μας να δυσφαλίσουμε τη συλλογή των δεδομένων. Επιδεινώθηκε η κατάσταση ή όχι. Για να απαντήσω και στις ε, δύο ερωτήσεις σχετικά με την Europol. Δεν έχω απάντηση, νομίζω ότι είναι και τα δύο. Ε, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη προσοχή από τα κράτη-μέλη απέναντι στον ε, κύκλο ευρωπαϊκής πολιτικής και εργάζεται περισσότερο για την εμπορία. Νομίζω ότι είναι επιτυχή αυτή η δραστηριότητα δηλαδή να συνεργάζονται τα κράτη-μέλη, γιατί πραγματικά συνειδητοποιούν ότι αυτό είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να προχωρήσουμε. Αλλά επίσης πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε και περισσότερα θύματα εμπορίας. Δεν έχω αριθμητικά στοιχεία, αλλά αυτό το λέω για να συνδεθώ και με τη δική σας ερώτηση. Νομίζω ότι σε καιρούς κρίσης η ευάλωτη κατάσταση κάποιων ατόμων αυξάνεται, επιδεινώνεται και βλέπουμε εδώ το θέμα της ισότητας και πού έγκυται αυτή η ισότητα. Στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται λόγος για τις αιτίες της εμπορίας ανθρώπων και μιλάει για κάποιους ανθρώπους που ζουν, παραδείγματος χάρη, σε περιοχές συγκρούσεων και είναι ευάλωτοι στο κοινωνικό αποκλεισμό. Ανισότητα μεταξύ ανδρών ε, βία που βασίζεται στο φύλλο. Όμω, αν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ένα κύριο παράγοντα, είναι η ευάλωτη κατάσταση ενός ατόπου σε συνδυασμό με την ανέχεια. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι πιο πιθανό όταν είναι ευάλωτοι άνθρωποι να είναι πιο εκτεθειμένοι και δεν είναι τόσο πιθανό κάποιος ε, από εμά ε, στην ε, αίθουσα εδώ θα ήταν αντικείμενο εμπορίας. Και ξέρετε, δεν αρπάζουν του ανθρώπου από κάποια άθεση. Πολλέ φορέ κάποιοι άνθρωποι ζητούν ευκαιρίε, ζητούν δουλειά και εδώ δεν μιλάμε για εργαζομένους χωρίς χαρτιά, μιλάμε για ανθρώπους που έκαναν αίτηση για ένα είδος δουλειάς ε, μέσω νόμιμων ή παράνομων ε, υπηρεσιών απασχόλησης και κατόπιν είναι αντικειμένο εμπορία. Έτσι λοιπόν δεν επιλέγουν τι συνθήκε εργασία του, δεν έχουν επιλογή ε, για τη δουλειά του, δεν μπορούν να διαφύγουν και του ε, κρατάνε είτε με απειλέ είτε με σωματική βία. Και αυτό συμβαίνει συνεχώ. Έχουμε πολύ μεγάλη τεκμηρίωση για αυτό το θέμα. Και όταν ε, μιλάμε για τις κυρίες αιτίε, τον ευάλωτο χαρακτήρα κτλ, πολλοί μας ρωτήσατε για το θέμα της ζήτησης θα έλεγα ότι αυτά είναι τα κύρια στοιχεία στα οποία επικεντρώνεται η Κομισιόν αυτή τη στιγμή και αυτό το κάνουμε με πολλούς τρόπους. Καταρχήν, η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ έρευνας ε, έχει ε, δημοσίευσει αυτό το διαγωνισμό για 12,5 εκατομμύρια έτσι ώστε τα πανεπιστήμια στην Ευρώπη να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες, να κατανοήσουμε την ζήτηση ε, για, τα, για θύματα της εμπορίας, Δεν μιλάμε για σεξουαλική είτε για έργαση και εκμετάλλευση. Πρέπει να καταρτήσουμε μία έκθεση σύμφωνα με την οδηγία αυτό το 2016 που να ε, προσεγγίζει το θέμα της πιθανής ποινικοποίηση των πελατών όταν ξέρουν αυτοί ότι πρόκειται για θύμα εμπορίας. Δηλαδή, δεν ε, απαντώ στην ευρύτερη ερώτησή σας για την πορνεία την εμπορία, αλλά όταν κάποιος γνωρίζει ότι χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ενός θύματος ε, να τιμωρείται. Τώρα, ε, αυτός δεν είναι στο μέσο που μπορεί να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν είναι σαφή ότι υπάρχει άμεσος σύνδεσμος μεταξύ πορνείας και εμπορίας. Και όπου υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος, πολλές φορές είναι ισχυρός αυτός ο σύνδεσμος όταν δούμε τα ποσοστά. Η Κομισιόν λοιπόν θα το παρακολουθήσει αυτό μέσω της οδηγίας. Η Κομισιόν επίσης ε, το Μάρτιο στη Νέα Υόρκη θα παρακολουθήσει μια διάσκεψη για τα δικαιώματα των γεγονών και εκεί θα συζητήσουμε το θέμα της διάστασης του φύλου και της εμπορίας γυναικών και κοριτσιών. Και, και εδώ λοιπόν ασχολούμαστε ενεργητικά. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε για την Κίνα και την Ιγυρία. Συγγνώμη, έχασα την ερώτηση. Όλα αυτά τα στοιχεία θα τα δείτε και στην έκθεση. Δεν θέλω τώρα να σας ε, δώσω περισσότερες πληροφορίες γιατί δεν μπορώ, αλλά πρόκειται για συγκεκριμένες χώρες. Ξέρετε, έχουμε κορίτσια και γυναίκες από την Ιγυρία σε ολόκληρη την Ένωση που είναι αντικείμενο σεξουαλική εκμετάλλευση και νομίζω ότι επικεντρώνεται σε τρει-τέσσερι χώρε. Βέβαια, αυτό θα δημοσιευτεί βάσει δεδομένων που θα δώσει το κράτη-μέλη. Το ίδιο και για την Κίνα για τα εγκληματικά δίκτυα, τα οργανωμένα δίκτυα. Δεν έχω εδώ την παράθεση της ε, Europol, δεν θα τη διαβάσω λοιπόν, αλλά Europol στην έκθεση 8 2011. Σαφέστατα αναφέρει συγκεκριμένες χώρες όπου υπάρχουν αυτά τα εγκληματικά δίκτυα, από όπου προέρχονται αυτοί οι έμποροι ανθρώπων και οι χώρε εντό Ένωση είναι το ένα. Οι χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση με τον κατάλογο που έχουμε στο έγγραφο προσανατολισμού δράση που δημοσιοποιήσαμε, θα δείτε ότι υπάρχει ισχυρό σύνδεσμο εκεί. Δεν είδαμε λοιπόν μόνο τον αριθμό των θυμάτων, αλλά και τους συνδέσμους με τα εγκληματικά δίκτυα. Και φυσικά αυτό έχει νόημα. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω για τη συνεργασία των κρατών μελών. κατανοώ ότι υπάρχει αυξανόμενη συνεργασία, γιατί υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση από τα κράτη-μέλη για περισσότερη συνεργασία. Δεν θα έλεγα ότι ισχύει με όλους. Υπάρχει πιο διμερής δουλειά. Μερικέ φορέ ενισχύεται αυτό και μέσω των κοινών ομάδων ε, και ω ένα βαθμό υπήρχε επιτυχία. Αλλά τώρα που στα μετά, όταν φτάνουμε στι διώξει. Είχαμε λοιπόν ένα πολύ καλό project εκτέθηκε ένα αριθμό δικτύων, αλλά όταν ε, φτάσαμε στι διώξει πόσο μάλλον καταδίκε ήταν πολύ χαμηλή η αριθμή. Τώρα επιφυλάσσομαι να πω γιατί έχουμε τόσο χαμηλό αριθμό, μέχρι να έχουμε την πλήρη μεταφορά τη οδηγία στο ιστορικό δίκαιο 6 Απριλίου φέτο. Στην οδηγία Υπάρχει μία διάταξη που αφορά πώς μπορούν να αυξήσουν τις διώξεις στα κράτη-μέλη και αναφερόμαστε και στις αυστηρές ποινές μέχρι 10 χρόνια κάθριξης για τους εμπόρους ατόμων. Ελπίζω λοιπόν ότι τον Απρίλιο θα μπορέσουμε να προκληθήσουμε πιο στενά τα γεγονότα. Σε ό,τι αφορά στις συστάσεις. Υπάρχει μια σειρά τομέων στη στρατηγική. Η δική μου σύσταση θα ήταν να δούμε το θέμα αυτό πιο συνολικά. Αν δούμε την απόφαση πλαίσιο του 2002, που αντικαταστάθηκε τώρα από την οδηγία, είχε μια πολύ ήπια προσέγγιση σε ό,τι αφορά την επιβολή του νόμου. Όμως η επιβολή του νόμου από μόνη της, δηλαδή αυτό που μας έχει δείξει η ιστορία, η δεκατής ιστορία, τη απόφαση πλαισίου και το τι μα είπαν τα κρατημέλη είναι ότι δεν ε, λειτουργήσει αρκετά καλά. Και πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στην πρόληψη, στην προστασία των θυμάτων και να βοηθήσουμε τα θύματα. Γιατί εν τέλει έχουμε πληροφορίες από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης ότι όταν πάρα πολλά θύματα επιστρέφουν στην πατρίδα τους, είτε εντός της Ένωσης είτε εκτός Ένωσης, τελικά καταλήγουν πάλι στα δίχτυα των εμπόρων. Έτσι λοιπόν πρέπει να διασφαλίσουμε ότι εντάσσονται και πάλι στην κοινωνία τα θύματα. Η στρατηγική της Κομισιόν από τον Ιούνιο του 2012 ακριβώ τονίζει την ανάγκη αυτή να διασφαλίσουμε μια πιο συντονισμένη προσέγγιση. Και φυσικά περιλαμβάνεται και μια σειρά δράσεις για τα κράτη, δράσεων για τα κράτη-μέλη. Έχουμε 40 δράσεις ε, σε ό,τι αφορά τις κλιματοοικονομικές έρευνες, ε, σε ό,τι αφορά τη δίωξη και σε τέτοια ζητήματα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μα υποστηρίζουν τα κράτη-μέλη στην προσπάθεια αυτή. Ελπίζω να απάντησα στι περισσότερε ερωτήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμεί πολύ για την σαφήνεια με την οποία απαντήσατε στις ερωτήσεις μας. Και σας ευχαριστούμε και για το έργο σας, που επίσης μας παρουσιάσατε σήμερα. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Τώρα περνάμε στο δεύτερο τμήμα εδώ θα δείτε κάποιον πιο νέο, τον κύριο Ταβάρης που θα αναλάβει την Προεδρία. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σε όλους. Κυρίως τον οξετιμό συνάδελφο Κίρκοπ που είχε την Προεδρία μέχρι τώρα. Περνάμε λοιπόν στη, στο δεύτερο τμήμα της σημερινής μας ακρόασης που έχει να κάνει με την συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες. Και πιο συγκεκριμένα παίρνουμε σαν παράδειγμα τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ρουσία. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ραούλ Ερνάντες η Σαγρέρα, που είναι από το Διεθνές Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών της Βαρκελόνης, που έχει ετοιμάσει μία μελέτη όσον αφορά την Ρωσία και τον κοινό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Έχετε 10 λεπτά και μετά φυσικά θα υπάρξουν και ερωτήσεις. Παρακαλώ κύριε Νάντης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πραγματικά είμαι ευγνώμων στην Επιτροπή σας που με κάλεσε να έρθω και να σας παρουσιάσω τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης μας όσον αφορά την Ρωσία και το κοινό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Την μελέτη αυτή την έκανα από κοινού με την δόκτωρα Όλγα Ποτέμκινα που είναι από το Ευρωπαϊκό από την ε, Ρωσική Ακαδημία Επιστημών και την ευχαριστώ πολύ βέβαια για τη συνεργασία. Η συνεργασία αυτή στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης εξετάζεται κυρίως από πλευράς έρευνας. Βέβαια έχει αρχίσει από το 1990. Στόχος πάντως της μελέτης μου εμένα είναι να υπογραμμίσουμε τι γίνεται σε αυτό το πολύ σημαντικό τομέα συνεργασίας τα τελευταία χρόνια, από τότε που άρχισε να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας δηλαδή, και τι αλλαγές και διορθώσεις έχουν γίνει τώρα που υπάρχει και η υπηρεσία η Ευρωπαϊκή Εξωτερικής Δράσης. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν τα κύρια συμπεράσματά μας, κάπως σύντομα, για να έχουμε χρόνο για ερωτήσεις και απαντήσεις. Η συνεργασία στο θέμα του οργανωμένου εγκλήματος με την Ρωσία, λέω ευθύ εξ αρχής, ότι δεν έχει προχωρήσει ιδιαίτερα. Θα επικεντρωθώ όμως παρόλα αυτά στην ε, όποια συνεργασία υπάρχει, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ακριβώς που σας ενδιαφέρει. Από πλευράς μεθοδολογίας, η μελέτη έχει συμπεριλάβει ε, τα αποτελέσματα διαφόρων συνεντεύξεων που είχαμε με διάφορους συθήνοντες από την Ρωσία, διευθυντές Ινστιτούτων, υπηρεσίες ε, εσωτερικών υποθέσεων και στην Ευρώπη βέβαια και στη Ρωσία. Θα σας παρουσιάσω πρώτα απ' όλα τους ε, στόχους και τα κύρια συμπεράσματα και μετά θα σας παρουσιάσω το κανονιστικό και το θεσμικό πλαίσιο της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας στον τομέα της ελευθερίας ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Και μετά το κυρίως τμήμα μου θα είναι οι διάφορες πολιτικές και η κατάσταση πραγμάτων για τους τρεις αυτούς τομείς. Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη. Θα σας πω πού έχει υπάρξει πρόοδος, για παράδειγμα όσον αφορά το χάρτη πορείας και τι έχει γίνει σε άλλες πολιτικές όπου έχουμε περιορισμένη πρόοδο. Και στο τέλος θα καταλήξω στα συμπεράσματά μας. Ποιοι είναι οι στόχοι λοιπόν της μελέτης αυτής. Πρώτα απ' όλα να αξιολογήσει την πρόοδο στην εφαρμογή του χάρτη πορείας όσον αφορά τον κοινό χώρο Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία. Δεύτερον, να αναλύσουμε τα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι υπάρχει αδυναμία στην συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ρωσία. Να ξέρετε ότι η μελέτη αυτή μου ζητήθηκε από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Πολλά μέλη της Επιτροπής αυτής κρίμε συμμετέχουν και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Έτσι δεν είναι, όπως επίσης και στην Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τη Ρωσία. Οπότε η Λίμπε όταν μας ζήτησε τη μελέτη αυτή τόνισε το θέμα της έλλειψης συνεργασίας με τη Ρωσία. Γιατί λοιπόν, ποιοι παράγοντες εξηγούν την έλλειψη αυτής της συνεργασίας. Αυτό θα σας παρουσιάσω και μετά θα κάνω μια αξιολόγηση της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πω και δύο λόγια όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας. Διότι τα διάφορα Ινστιτούτα ή οργανώσεις και τα λοιπά που συμμετέχουν στη συνεργασία στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης επηρεάζουν και τα αποτελέσματα. Τώρα σας είπα ήδη ότι ο χάρτης πορείας δεν εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο στον τομέα της ε, ασφάλειας, για παράδειγμα, με την, με την επανεισδοχή που δεν ε, προχωράει αρκετά ή με τα θέματα ελευθέρωσης θεωρήσεων. Ένα άλλο συμπέρασμά μας είναι ότι υπάρχει έλλειμμα και στην αμοιβή εμπιστοσύνη σε πολιτικό επίπεδο και ότι ο τρόπος που χρησιμοποιεί την αιρεσιμότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως να βρίσκεται πίσω ακριβώς από την έλλειψη αυτή αμοιβαίας εμπιστοσύνη. Και τι εννοώ, εννοώ ότι υπάρχουν ε, όλο και περισσότερες επαφές μεταξύ εμπειρογνωμόνων εκατέρωθεν και εμείς πιστεύουμε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να ενισχυθεί στο μέλλον η συνεργασία με τη Ρωσία. Τώρα πολύ γρήγορα θα αναφερθώ στο κανονιστικό πλαίσιο. Να κάποιες έννοιες που είναι αναγκαίες για να καταλάβουμε από πού ερχόμαστε και πού πάμε όσον αφορά τη συνεργασία μας με τη Ρωσία στους τομείς αυτούς. Ξέρετε ότι το δεσμευτικό πλαίσιο της συνεργασίας είναι η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας που άρχισε να ισχύει το 1997 Βέβαια υπήρχε ένα πολύ ασαφές κεφάλαιο, το κεφάλαιο 8, όσον ε, αφορά τη συνεργασία σε θέματα παράνομων δραστηριοτήτων. Μετά είχαμε μια νέα βάση συμφωνίας για να ρυθμιστούν γενικότερα τα θέματα ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Τώρα υπάρχουν ε, διαπραγματεύσεις που θα αντικαταστήσει η νέα συμφωνία εκείνη της εταιρική σχέσης και συνεργασίας. Όσον αφορά τώρα το μη δεσμευτικό πλαίσιο, το 2003 με τη διάσκεψη κορυφής ε, στο Σιντ Πέτερσβουρκ τέθηκε η μερίσια διάταξη για συνεργασία που διευκρινίστηκε παρετέρω με το χάρτη πορείας που εγκρίθηκε στη συνέχεια και άρχισε να ισχύει από το 2005. Είναι μια πολιτική ατζέντα. Είναι αυτή που έχουμε και βάσει αυτής πορευόμαστε. Στη συνέχεια έχουμε το πρόγραμμα ε, της Στοκόλμης που ορίζει την Ρωσία ως εταίρος στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Και όπως είπα και στην αρχή, με τη συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύεται ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εξωτερική δράση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του για διεθνείς συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα θα περάσω στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την συνεργασία μας με την Ρωσία στους τομείς αυτούς. Συναντήσεις, διαπραγματεύσεις γίνονται στα πλαίσια του μόνιμου Συμβουλίου Εταιρικής Σχέσης, Permanent Partnership Council. Αν συγκρίνουμε αυτό το PPC, αυτό το ομώνυμο Συμβούλιο Εταιρικής Σχέσης, <clears throat> με τις υποεπιτροπές οι οποίες λειτουργούν για την ε, συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις γείτονες χώρες, οι υποεπιτροπές αυτές είναι πολύ περισσότερο δομημένες. Και υπάρχει μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα μέσα σε αυτές από υπουργεία, είτε εσωτερικών είτε γιατί Η προσώπευση είναι καλύτερη σε αυτές. Το μόνο που θέλω εδώ να υπογραμμίσω είναι ότι οι υποεπιτροπές είναι ένας ε, πιο ευνοϊκός χώρος για τις επραγματεύσεις από το Συμβούλιο για την συνεργασία μας αυτή. Γι' αυτό και μόνο για πολύ συγκεκριμένες ε, πολιτικές, για τις θεωρήσεις, για παράδειγμα, ή για άλλα θέματα συνεδριάζει το Συμβούλιο αυτό. Και αυτό που λέμε στην μελέτη μας είναι ότι τέτοιες συναντήσεις λαμβάνουν χώρα γενικά για όλες τις πολιτικές, ορισμένες τουλάχιστον, γενικά για τη συνεργασία στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Στην τελευταία μάλιστα συνεδρίαση είπαν ότι μια φορά το χρόνο πρέπει να συναντιόνται και να καλύπτουν όλους τους τομείς. Τώρα έρχομαι στην πρόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θα συντονίσει καλύτερα την εξωτερική της δράση στους τομείς ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Και εδώ έχουμε την ε, ανάμειξη και τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Γενική Διεύθυνση Home, η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς που ασχολούνται με την ε, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη έχουν παίξει ζωτική σημασία ρόλο στην εφαρμογή του χάρτη πορείας. Η Frontex, η Europol, η Sepol, Όλοι αυτοί έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Και με την συνθήκη της Λισαβόνας βλέπουμε ότι έχουμε νέες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από αυτήν την εισαγωγή για το πού βρισκόμαστε, θα έρθω στην ε, αξιολόγηση των διάφορων πολιτικών. Ξεκινώντα με εκείνε τι οποίε έχει επιτευχθεί πραγματική πρόοδο. Πρώτα απ' όλα η Συμφωνία Επανεισδοχή. Εδώ έχει εφαρμοστεί επιτυχώς από το 2007 και μετά δεν υπάρχουν ε, σοβαρά προβλήματα και διαμαρτυρίες από τη μία την άλλη πλευρά. Φυσικά και τα κράτη-μέλη συμμετέχουν στην εφαρμογή της συμφωνίας αυτής. Η μόνη δυσκολία που έχουμε εντοπίσει είναι αυτή που έχει να κάνει με τον εντοπισμό της υπηκότητας των ανθρώπων που περνάνε από τη Ρωσία, χωρίς όμως να ξεκινάνε από τη Ρωσία, περνάνε από την Ρωσία για να καταλήξουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως transit. Δεύτερο θέμα, διαχείριση συνόρων. Υπάρχει συνεργασία ε, μεταξύ της Frontex και της αντίστοιχης υπηρεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η συμφωνία αυτή έχει αρχίσει από το 2006. Πρόκειται για την οικοδόμηση ικανοτήτων, υπάρχουν τέτοια προγράμματα όσον αφορά την ε, παράνομη μετανάστευση. Υπάρχει επίσης και κάτι όσον αφορά Όσον αφορά την οριοθέτηση συνόρων, υπάρχει συμφωνία με την Λετωνία και την Λιθουανία και γίνονται, μάλλον και ολοκληρώθηκαν και διαπραγματεύσεις με την Εστονία. Έρχομαι τώρα σε άλλες πολιτικές και θα δείτε ότι είναι περισσότερες από αυτές που σας είπα ήδη ότι έχει υπάρξει πρόοδος. Υπάρχουν άλλες λοιπόν πολιτικές όπου έχουμε λιγότερη πρόοδο. Το θέμα της ελευθέρωσης <clears throat> του καθεστώτος θεωρήσεων, δηλαδή η κατάργηση των θεωρήσεων ε, που απαιτούνται βάση Σέγγεν από τους ε, Ρώσους και αντίστοιχα που ζητάει η Ρωσία από τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι πολύ σημαντικός τομέας αυτός. Διότι στην διαδικασία αυτή εμπλέκονται όλες οι πολιτικές που έχουν να κάνουν με την ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη. Μιλάμε για ένα κοινό χώρο, πρέπει εδώ να οριστούν τεχνικές προδιαγραφές και βλέπουμε ότι χρειάζεται συνεργασία σε πράγματα που έχουν να κάνουν είτε με την ασφάλεια των γράφων, δηλαδή βιομετρικά διαβατήρια, έλεγχο τη ε, παράτυπη μετανάστευση, πώς δηλαδή θα εφαρμόζεται σωστά η Συμφωνία επανεισδοχή, τίθενται θέματα δημόσιας τάξης και προστασίας, πολύ σημαντικά, αλλά λάβουμε υπόψη μας το οργανωμένο έγκλημα, εδώ έχουμε να κάνουμε με θέματα επιβολής του νόμου και υπάρχει και κάτι που είναι πιο ασαφές, είναι οι εξωτερικές σχέσεις και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Όταν μιλήσω για τη συνεργασία μας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα επανέλθω σε αυτό. Πάντως, η Ρωσία έχει συμφωνήσει ότι εφόσον υπάρξουν έτοιμες όλες αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές, τότε θα υπάρξει το επόμενο βήμα που θα οδηγήσει στην κατάργηση των θεωρήσεων. Ποια είναι η κατάσταση πραγμάτων τώρα όσον αφορά την εφαρμογή όλων αυτών. Η Ρωσία βέβαια λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αρκεί να πάρει την πολιτική απόφαση να καταργήσει και ότι αυτό αποτελεί προτεραιότητα για τη Ρωσία. Έτσι λένε οι Ρώσοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της τονίζει την τεχνική πτυχή, δηλαδή πώς θα εφαρμοστούν όλε οι προϋποθέσεις που πρέπει να εφαρμοστούν προηγουμένως. Άρα η προσέγγιση είναι διαφορετική ε, κατέρωθεν. όσον αφορά την ε, διαδικασία ελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων. Τώρα υπάρχει και η συμφωνία για την διευκόλυνση θεωρήσεων του 2007. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει πιο απλές διαδικασίες για ορισμένες κατηγορίες ατόμων που ζητούν θεώρηση. Αυτή είναι μια συμφωνία που ισχύει τώρα. Πρέπει όμως να τροποποιηθεί και να αντικατασταθεί από μια νέα συμφωνία, που χρειάζεται βέβαια τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα προσαρμόζει τις προδιαγραφές στον κώδικα θεωρήσεων που εγκρίθηκε το 2009. Και εδώ, επειδή δεν υπάρχει αμοιβή εμπιστοσύνη, όπως είπαμε πριν, μεταξύ των δύο πλευρών, όσον αφορά την εφαρμογή του συστήματος θεωρήσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να συμπεριληφθούν αυτοί που έχουν υπηρεσιακά διαβατήρια στη Νέα Συμφωνία, η Ρωσία μετά από αυτό αντέδρασε αρνητικά και κατήργησε τη πρόβλεψη αυτή ειδικών κατηγοριών, για παράδειγμα πληρωμάτων, που έχεραν από αυτή την ε, συμφωνία διευκολύσεων θεωρήσεων. Δηλαδή η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσματα. Υπάρχει τώρα και η συμφωνία για το Καλίνιγκραντ. Εδώ έχουμε συμφωνία για διευκόλυνση της επικοινωνίας των κοινωνιών που ζουν εκατέρωθεν των συνόρων αυτών. Το Καλίνιγκραντ ακριβώς επειδή πρόκειται για θύλακα, έχει ειδική ρύθμιση από την Πολωνία. Όλη η επαρχία του Όμπλας καλύπτεται από την συμφωνία και υπάρχει συμφωνία και με την Ορβηγία. Ω δεδεμένο κράτος με το Σέγγεν, η Νορβηγία μπορεί επίσης να συμμετέχει στην ρύθμιση αυτή. Αλλά εκκρεμεί ακόμα συμφωνία με τη Λιθουανία. Συνεργασία τώρα στον τομέα των ναρκωτικών. Εδώ έχουμε άλλη μια ευρωπαϊκή υπηρεσία, εκείνη του ελέγχου του Κέντρου για τα Ναρκωτικά και υπάρχει και από τη Ρωσία μια αντίστοιχη υπηρεσία. Έχει ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των δύο ε, με μια συμφωνία που προβλέπεται για το 2013. Για τα πρόδρομα ναρκωτικά θα υπογράψουν μια συμφωνία λοιπόν οι δύο πλευρές το 2013. Έχουμε αναλύσει στην ε, ε, μελέτη μας τον διάλογο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Είναι κάτι που έχει ξεκινήσει από το 2011. Είναι μια θεματική συνεργασία που λαμβάνει χώρα για την νόμιμη μετανάστευση, το άσυλο, την ένταξη των μεταναστών. Όλοι οι ειδικοί και πυρογνώμονες και αξιωματούχοι με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή μας είπαν ότι τώρα πρέπει να περάσουμε στο επιχειρησιακό στάδιο. Στο στάδιο εκείνο δηλαδή που δεν θα γίνεται μόνο ανταλλαγή απόψεων, αλλά θα προχωρήσουμε περισσότερο και σε εφαρμογή. Συνεργασία τώρα για το διασυνοριακό έγκλημα. Για την καταπολέμησή του βέβαια. Δεν έχει προχωρήσει πολύ μεταξύ των δύο πλευρών. Υπάρχει όμως συνεργασία. Και οι κύριες δομές ή κύρια μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας είναι υπογραφή μιας συμφωνία συνεργασία μεταξύ Europol και Ρωσία το 2003 που προβλέπει ανταλλαγή πληροφοριών, βέλτιστες πρακτικές, μελέτες, επισκέψεις. Όπως επίσης προβλέπει και τη δημιουργία ενός ε, ρωσικού σημείου επαφής με την Europol. Έπειτα υπάρχει και το σχέδιο πρωτοκόλλου ανάμεσα στη Σεπόλο και την Ακαδημία Διαχείρισης του Ρωσικού Υπουργείου Εσωτερικών. Έχει υπογραφεί όμως τελικά αυτή. Και υπάρχει και το κυβερνό έγκλημα. Εδώ πρέπει να οριστεί καλύτερα η ασφάλεια από το κυβέρνο έγκλημα. Γίνονται συζητήσεις αυτή την εποχή για την συνεργασία όσον αφορά τον κυβερνοχώρο μεταξύ των δύο πλευρών. Η Ρωσία όμως δεν θέλησε να υιοθετήσει την ε, σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το κυβερνό έγκλημα και αυτό όπως καταλαβαίνετε εμποδίζει τις εξελίξεις. Κάτι άλλο σημαντικό είναι οι συμφωνίες για συνεργασία με την Europol και την Eurojust δεν έχουν προχωρήσει. Δεν συμμορφώνεται η Ρωσία με τις προδιαγραφές και αυτό είναι που εμποδίζει και την σύναψη συμφωνίας για το τρόπο εργασίας, τη συνεργασία. Η Ρωσία όμως κύρωσε την, ε, μάλλον όχι βρίσκει ακόμα από πλευρά της Ρωσίας η πρόταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την σύμβαση ποινικού δικαίου όσον αφορά την διαφθορά. Τι άλλες εξελίξεις τώρα αξίζει να αναφέρουμε. Όσον αφορά την διαφθορά. Εδώ έχει υπάρξει υπογραφή το 2007. Έρχομαι τώρα στη συνεργασία όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Η βάση είναι η βάση μάλλον για τη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών όσον αφορά την ελευθερία, την ασφάλεια και την δικαιοσύνη. Όμως, ε, κατέρωθεν υπάρχει μια αρνητική αξιολόγηση της κατάστασης. Από το 2005 έχουμε διαβουλεύσεις δύο φορές το χρόνο, στις Βρυξέλλες πάντα, που θεωρούμε ότι έχουν ελάχιστα αποτελέσματα. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε ενίσχυση των διαβουλεύσεων αυτών, ζήτησε πιο ενεργό συμμετοχή και ζήτησε να γίνονται εκ περιτροπής μια φορά στις Βρυξέλλες και μια φορά στη Μόσχα οι διαβουλεύσεις αυτές. Δημιουργήθηκε και ένα φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών το 2011 που μπορεί να συμμετέχει επίσης. Θέλω σε αυτό το σημείο να υπογραμμίσω τα συμπεράσματα του τελευταίου μόνιμου Συμβουλίου συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση Ρωσία που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο μας πέρασε στη Λευκοσία. Για πρώτη φορά αποφάσισαν οι δύο πλευρές να αναφερθούν στην αρχή της ανεξαρτησία της δικαιοσύνη. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ανεξάρτητη δικαιοσύνη, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα στοιχείο κλειδί για την απρόσκοπτη επιβολή του νόμου και για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο. Οι δύο πλευρέ επίση αναφέρθηκαν στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτου δικαίου, χωρί όμω να αναφερθούν στην πρόθεση τη δημοκρατία στα συμπεράσματά του, στα συμπεράσματα αυτού του μόνιμου συμβουλίου που σα είπα το Οκτωβρίου που μα πέρασε. Όταν αναφέρθηκα στη διαδικασία για, την, για τις θεωρήσεις, είπα Πώ ε, εμπλέκεται και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και από τι δύο πλευρές πάντως υπάρχει μια δέσμευση συνεργασία στα ανθρώπινα δικαιώματα. όμω δεν αναφέρεται σε τι βαθμό θα γίνεται αυτό. Δηλαδή αυτή η δέσμευση για συνεργασία στην πράξη τι σημαίνει. Αν προσπαθήσουμε να κάνουμε μια αναλογία της κατάστασης στη Ρωσία, όπως στην Ουκρανία, τη Μολδαβία για τις θεωρήσεις, Εκεί είχαμε πει συγκεκριμένα ε, ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις. Αυτό όμως δεν αναφέρεται στη συνεργασία με την Ρωσία και μάλιστα είναι κατά από ό,τι φαίνεται η Ρωσία μιας συνεργασίας για νομοθεσία που να ε, καταργεί τις διακρίσεις. Συμπεράσματα. Και έχω τηρήσει το χρόνο μου νομίζω. Θέλω εδώ να συνδέσω λιγάκι τα ανθρώπινα δικαιώματα με την αβεβαιότητα που επικρατεί. Ένα από τα στοιχεία που θέλω να υπογραμμίσω εδώ είναι την έλλειψη διαφάνειας όταν γίνονται διαπραγματεύσεις σε θέματα ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών. Και γιατί, γιατί οι δύο πλευρές δεν είναι διατεθειμένες να φέρουν στη δημοσιότητα τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν. Για παράδειγμα, τα διάφορα βήματα τα οποία έχουν αναλυθεί για την ελευθέρωση ε, των θεωρήσεων, την κατάργησή τους, δεν έχουν ε, δημοσιοποιηθεί. τι έχει εφαρμοστεί κάθε φορά για να μπορεί κανείς να τα παρακολουθήσει αυτά. Δεν υπάρχει αρκετή διαφάνεια, δηλαδή ούτε είναι γνωστά τα διάφορα έγγραφα ε, τα οποία ετοιμάζονται και εκπονούνται κατά διάρκεια των ε, διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, πρώτο συμπέρασμα. Δεν εφαρμόζεται ικανοποιητικά ο χάρτης πορείας. Στο διάλογο για την κατάρχηση των θεωρήσεων τα περισσότερα μέτρα έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των συνόρων, για παράδειγμα. Θέματα που έχουν να κάνουν με την ελευθερία είναι πλήρως απόντα. Θα ήθελα να σκεφτείτε λιγάκι ποιος θα ήταν ο ορισμός της ελευθερίας, των θεμάτων που έχουν να κάνουν με την ελευθερία. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ήδη εγκρίνει διάφορα μέτρα για την νόμιμη μετανάστευση. Έχουμε ολόκληρο πακέτο, έχουμε την οδηγία για την μπλε κάρτα. για τους εποχιακούς ε, εργαζόμενους κλπ. Όλα αυτά είναι μέτρα νόμιμα που έχουν ήδη εγκριθεί, που αποτελούν μέρος της ημερήσιας διάταξης και έχουν μια εξωτερική διάσταση και θα έπρεπε να εφαρμόζονται από κοινού με τρίτες χώρες. Όταν λοιπόν συζητάμε την ατζέντα ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης με τη Ρωσία ή και με άλλες χώρες, θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται και τέτοια θέματα ελευθερία, ελεύθερη διακίνηση είναι πράγματα τα οποία δεν θα πρέπει να μας περιορίζουν στις θεωρήσεις, αλλά να έχουν να κάνουν και με άλλες μορφές μετακίνησης. Γιατί τώρα, ποια άλλη λόγοι υπάρχουν που δεν υπάρχει πρόοδος. Έλλειψη εμπιστοσύνη είπαμε. Όχι σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, το θέμα της ρεσιμότητας, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για προοπτική. Θέλει πάντα να υπάρχει μια συμμετρία, να φαίνεται δηλαδή ότι είναι επίσης όρις οι δύο πλευρές. Είπαμε ότι θέλουμε περισσότερες επαφές και ενίσχυση της εμπιστοσύνης. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη μέθοδος για να υπάρξει κάποια πρόοδος στη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω τώρα τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ερνάντες Σαγρέρα. Και τώρα θα δώσω το λόγο για τις ερωτήσεις. Να ξεκινήσουμε με τους συντονιστές και γιατί ξέρω ότι βιάζεται, κυρία Φαγιάν, όχι. ο κύριος Μποργέτσιο. Κύριε Νιντονταν και εσείς. Να ξεκινήσουμε τον κύριο Μποργέτσιο. Κατόπιν κύριε Μορβάη και κύριος Νιντονταν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Τα θέματα που θίξατε είναι όλα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Εγώ θα επικεντρωθώ σε μια πτυχή που αναδύθηκε και που με ενδιαφέρει και το παρακολουθώ με ιδιαίτερη προσοχή θέμα που τα θέματα που σχετίζονται με το ξεπλήμα βρωμικού χρήματο και την παράνομη χρηματοδότηση. Κατά τη διάρκεια των εργασιών μας στις εκράσεις ε, είδαμε πάρα πολλά στοιχεία που μας οδηγούν στο να σκεφτούμε ότι υπάρχει μια μεγάλη κυκλοφορία αμφίβολων κεφαλαίων ε, προέλευσης εγκληματικής από τη Ρωσία προς τις ευρωπαϊκές χώρες. Και σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τύπο υπάρχει και μία είδηση για κατάθεση 26 ε, δισεκατομμυρίων ευρώ ρωσικής προέλευσης σε κυπριακές τράπεζες. Οι επαφές, οι συνεδριάσεις που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας για τα θέματα αυτά. Έχουν μπορέσει να προσεγγίσουν αυτές τις σημαντικές πτυχές. Γιατί η είδηση που κυκλοφορεί στο χρηματοοικονομικό κλάδο είναι ότι ε, υπάρχουν ε, πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις ρωσικών κεφαλαίων ε, και μιλάμε για πρόσωπα που έχουν πολύ μεγάλα ποσά, των οποίων δεν γνωρίζουμε ακριβώς την προέλευση. Μήπως σκέφτεστε να υπάρξει μία δράση αντιλαγής πληροφοριών και συνεργασίας για αυτό τον ευαίσθητο τομέα. now, Mrs. Η κυρία Μόρβα, ευχαριστώ. Από ό,τι κατάλαβα και από τον τίτλο της έκθεσης, Μιλάμε για συνεργασία με τη Ρωσία της Ένωσης πάνω στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και χαίρομαι που είπατε τέλος για μια αμοιβαιότητα και τον γνήσιο, τον πραγματικό χαρακτήρα της συνεργασίας. Είμαι ευαίσθητη για το θέμα γιατί είμαι Ανατολικοευρωπαία και μετά τη δημοκρατική μετάβαση περάσαμε μια περίοδο που η δυτική ήρθαν στη χώρα μου και μας ε, έβγαζαν λόγους για το τι θα έπρεπε να κάνουμε. Ίσως είμαι υπερβολικά ευαίσθητη, αλλά πρόσεξα ότι μιλήσατε για ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία, αλλά υπάρχουν μεγάλα προβλήματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν πάτε στο YouTube και γράψετε ας πούμε ε, παναυσότητα της αστυνομία της Ένωσης θα δείτε αποτρόπαια πράγματα σχετικά με τη βαναυσότητα της αστυνομία στην Ισπανία, την Ουγγαρία το 2006 και Βέβαια, πολλές φορές είναι πολύ βίαιοι απέναντι στους διαδηλωτές για τα μέτρα λιτότητας κλπ. Οπότε δεν κατάλαβα τι έχει, τι, αντικείμενο έχει αυτή η συνεργασία. Θέλουμε να τις πούμε της Ρωσίας τι να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ίδιο αφορά και τις διακρίσεις. Δηλαδή, τι έχει να κάνει η διάκριση με τα συγκεκριμένα θέματα. Μην με παρεξηγήσετε. Βεβαίως και είμαι μεγάλη υπέρμαχος το, ε, ε, της πολιτικής κατά των διακρίσεων. Σε ό,τι αφορά τη Ρωσία όμως, και εμείς έχουμε να μάθουμε ως δυτικοί από την ε, Ρωσία όταν μιλάμε για κατάργηση διακρίσεων στο χώρο εργασίας, τη σωστή συμπεριφορά στο χώρο εργασίας, ε, τη δημόσια ζωή. Μπορείτε να με διαφωτίσετε για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτούς τους δύο τομείς. Όταν μιλάμε για συγκεκριμένες ε, παραβιάσεις, ε, μπορώ να συμφωνήσω, αλλά για τις διακρίσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικότερα, τι, τι θα ε, πείτε στη Ρωσία και πώς συναρτώνται όλα αυτά με τα συγκεκριμένα προγράμματα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Ο κύριος Νιούτον Τζαν, ευχαριστώ πολύ. Πολύ εντυπωσιακή και συνεκτική περιγραφή όλη της κατάστασης. Μου έκανε εντύπωση ακούγοντά σα ότι υπάρχει ένα πολύ καλό πλαίσιο, αλλά δεν δουλεύει στην πράξη από ό,τι κατάλαβα, λόγω τη έλλειψη πολιτική βούληση, όχι από τη δική μα την πλευρά μάλλον, αλλά από την πλευρά τη Ρωσία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένα τομέα που μελέτησα αφορά τη λαθρεμπορία τσιγάρων από Ρωσία, Λευκορωσία, Ουκρανία. Το Καλίνιγκραντε είναι επίσης ιδεώδης ε, τόπος για να μπαίνουν τσιγάρα από εκεί, καλές μάρκες, ρωσικές μάρκες, ανατολικοευρωπαϊκές μάρκες και έχω την εντύπωση, παρόλο που κάνατε πολλή δουλειά για τη δημιουργία αυτού του πλαισίου, παρόλα αυτά δεν λειτουργεί αποτελεσματικά. Ή θα μου απαντήσετε ότι δουλεύει, λειτουργεί καλύτερα από ό,τι έχω την εντύπωση εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Να προσθέσω κι εγώ κάποιες ερωτήσεις πρώτη αφορά το οικονομικό έγκλημα και τη χρήση ως διάβλων των ε, κρατών μελών της Ένωσης ε, που ε, δρούν ως μέρη ξεπλήματος χρήματος που κερδίθηκε στη Ρωσία ή προέρχεται από τη Ρωσία. Και πώς επιστρέφουν πάλι αυτά τα χρήματα. Διάβασα πρόσφατα ότι η Κύπρος ήταν η ο τρίτος σε μέγεθος επενδύτη επενδυτής σε άμεσες επενδύσεις. Αυτό είναι περίεργο. Γιατί είναι η μισή Ιρλανδία. Παρόλο που δραστηριοποιούνται και οι μεγάλοι οικονομικοί όμιλοι. Εντυπωσιάζει λοιπόν το γεγονός ότι είναι τρίτος σε μέγεθος επενδυτής χρησιμοποιείται λοιπόν η Κύπρος ε, ως ε, κύκλωμα ξεπλήματος ε, χρήματος από τη Ρωσία που επιστρέφει στη Ρωσία. Εμείς τι εργαλεία έχουμε στη φαρέτρα μας για να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Και τώρα βέβαια δημιουργείται και μια τραπεζική ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να υπάρχει κεντρική εποπτεία των τραπεζών. Τώρα για το Συμβούλιο της Ευρώπης και αν ο ρόλος του βοήθησε ή όχι μέχρι τώρα για να ε, αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Γιατί η Ρωσία δεν, ε, δεν έχει προοπτική να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, υπάρχουν διμερείς σχέσεις και υπάρχει και ένας ε, οργανισμός ε, αιγίδα που είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης και μπορεί να βάλει μέσα από διαφορετικό πρίσμα τη συνεργασία. Τέλος, θέλω να μου πείτε αν η εντύπωση μου είναι σωστή, ότι έχουμε πολλά εργαλεία, αλλά πάμε να βάλουμε κύβους μέσα σε στρογγυλές σοπές. Και η περιορισμένη πρόοδος είναι κάτι αντικειμενικό ή τελικά διαχρονικά παρατηρήθηκε περισσότερη παλινδρόμηση παρά πρόοδος. Ορίστε. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής, ευχαριστώ πολύ που θέσατε όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί μου δίνουν την ευκαιρία να εξηγήσω περισσότερο τα απορίσματα της μελέτης. Τώρα, για το ξέπλυμα του χρήματος, ήθελα να θέσω το θέμα, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει μέχρι τώρα συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας μέσα στις επίσημες δομές. Από ό,τι ξέρω, το ξέπλυμα χρήματος δεν ετέθη ποτέ στο μόνιμο Συμβούλιο Εταιρική Σχέσης και στις συνεδριάσεις του και η Ένωση προσπάθησε να θέσει το θέμα, να γίνει ανταλλαγή απόψεων επ' αυτού, αλλά δεν είναι ένα θέμα όπου υπάρχει συνεργασία. Δεν τη βλέπουμε αφού δεν υπάρχει. Νομίζω ότι τα βασικά μέσα που μπορεί να αλλάξουν την κατάσταση αυτή θα είναι η θέσπιση ε, ρυθμίσεων συνεργασίας Europol-Eurojust όταν εγκριθεί το κείμενο αυτό το ξέπλυμα του χρήματος θα το καταπιαστούν και η συνεργασία θα μπορούσε να έχει αντικειμενική βελτίωση και τα θέματα θα τα ε, εξέταζαν σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, σχετικά με τα σχόλιά σας, καταλαβαίνω τις απόψεις σας. Στην έκθεση ακολουθούμε την ίδια γραμμή πλεύσης όπως και εσείς. Στο τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα στο θέμα των διακρίσεων, στο θέμα της καταπολέμησης των διακρίσεων, στρατηγικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση το καλύτερο θα ήταν να δεχτεί ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα προβλήματά της στον τομέα αυτό. Τώρα η αξιολόγηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ένθεν και κήθεν και από τις δύο πλευρές, γιατί η Ρωσία το βλέπει σε πολιτικό επίπεδο και επικρίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της κατάστασης των ρωσικών μειονοτήτων σε Λετωνία-Εσθονία. Αλλά και ε, γι' αυτό μιλάμε για κοινωνικοποίηση και όχι η αιρεσιμότητα. Η Ρωσία είναι πολύ ευαίσθητη απέναντι σε οποιαδήποτε επίκριση για τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί έγιναν πολλές επικρίσεις από ανεξάρτητους οργανισμούς, οργανώσεις, αλλά θέλει και αυτοκριτική. Θέλουμε λοιπόν λέμε στην έκθεση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη Ρωσία σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, όχι με τρόπο πατερναλιστικό. Οπότε ε, πραγματικά κατανοούμε και ως ένα βαθμό ασπαζόμεθα αυτά που είπατε. Τώρα, για τη λαθρεμπορία, ιδιαίτερα ο καθεστώς του Καλίνιγκραντ και τη λαθρεμπορία, πάλι όπως το ξέπλυμα χρήματος, και από ό,τι γνωρίζω, το θέμα της λαθρεμπορίας δεν έχει τεθεί σε αυτές τις ε, θεωρητικές ε, ε, ανταλλαγές απόψεων για το οργανωμένο έγκλημα. Αλλά η ανατροφοδότηση που παίρνω από την υλοποίηση της συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Πολωνίας, ιδιαίτερα στα σύνορα με το Καλίνιγκραντ δείχνει ότι δεν υπάρχει αύξηση της λαθρεμπορίας μεταξύ των δύο. Δεν θα μπορούσα να σας δώσω αριθμητικά στοιχεία, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι σοβαρό θέμα. Προφανώς και πρέπει να μας απασχολήσει γιατί μιλάμε για εγκληματική δραστηριότητα, αλλά δεν είναι ένα ε, πρόβλημα που ε, επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια. Τέλος, ε, για να απαντήσω στα δικά σας σχόλια, κύριε Πρόεδρε, για το Συμβούλιο της Ευρώπης και αν είναι χρήσιμος ο ρόλος του ή όχι, νομίζω ότι είναι χρησιμότατος ε, γιατί υπενθυμίζει στη Ρωσία ότι ως μέλος ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης θα πρέπει να προβεί στην εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων. Ε, πρέπει δηλαδή και να θεσπίσει νομοθεσία και να την εφαρμόσει. Αυτό ε, έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά. Γιατί δεν πρόκειται εδώ για ενωσιακά πρότυπα, αλλά πρότυπα που έχει ασπαστεί και ε, η ίδια η χώρα. Αξιοποιείται λοιπόν το καθεστώς του μέλου... στο Συμβούλιο της Ευρώπης για να ενθαρρυνθεί η Ρωσία να ε, εφαρμόσει κάποια πρότυπα. Είναι πολύ καλό. Τώρα, αν υπήρξε πιστοχώρηση ή πρόοδος στο νοδικό χάρτη, ε, νομίζω ότι παρόλα αυτά που σας είπα επιτελέστηκε πρόοδος. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ε, παρόλο που η Ρωσία δεν είναι στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία, παρόλο που η Ρωσία συχνά θεωρείται ως μια ειδική περίπτωση χώρας ε, με την οποία διαπραγματευόμαστε και είναι δύσκολο να γίνονται διαπραγματεύσεις και να επιτυγχάνονται συμφωνίες. Και η Συμφωνία Επανεισδοχής και της Διευκόλυνσης των Θεωρήσεων, ε, οι δύο συμφωνίες ε, πρώτα συμφωνήθηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή με τη Ρωσία σχέση με άλλε χώρε επίση. Οι ε, συνθήκες με τη Frontex πρώτα εφαρμόστηκαν με την Ρωσία, οπότε βλέπουμε εδώ συνεργασία. Υπάρχουν προφανώς πολλές προκλήσεις και αυτό είναι ο σκοπός της μελέτης, να ε, δώσει μια σύγχρονη εικόνα της κατάστασης και να εντοπίσει τα στοιχεία εκείνα που αποτελούν προσκόμματα για τη συνεργασία. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες διευκρινήσεις από τους παρισταμένους. Αν όχι, ευχαριστούμε για αυτή την εντυπωσιακή ανασκόπηση των προκλήσεων και στις σύνθετες σχέσεις Ρωσίας-Ένωσης. Ευχαριστώ άλλη μια φορά. Α, θα, το έχουμε, θα συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα μας σύντομα. Και πάμε τώρα στην επόμενη, τρίτη ενότητα, που αφορά την ε, διακρατική εγκληματικότητα. Οργανωμένο, το, διακρατικό οργανωμένο έγκλημα και τις οικονομικές διασυνδέσεις με την πειρατεία. Και το παράδειγμα της πειρατείας ε, έξω από τις ακτές της Σομαλίας. Και θα έχουμε μαζί μας τον αντιστράτηγο Τον Βαν Ως από το επιτελείο της ε, Ένωσης, τη Γενική Διεύθυνση και θα μιλήσει για την ε, επιχείρηση Αταλάντα για την καταπολέμηση της πειρατείας στην Σομαλία και της, ε, το διακρατικό οργανωμένο έγκλημα με τις οικονομικές του διακλαδώσεις. Έχουμε και τον κύριο Πέτερ Κώστερ, περιμένουμε τον κύριο Φανός. Ο κύριος Κώστερ είναι υπεύθυνο των επιχειρήσεων, επικεφαλής των επιχειρήσεων κατά της τρομοκρατίας και του οικονομικού εγκλήματος στην Europol και θα μας μιλήσει για την διασύνδεση πειρατείας και διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος και την πρόληψη, εντοπισμό και την ε, κατάσχεση. Thank Mr. General, well, I will give you the floor. Κύριε Αντιστράτηγε, θα σας δώσω το λόγο. Έχετε περίπου 15 λεπτά για την παρουσίασή σας και κατόπιν θα ακούσουμε τον κύριο Κώστερς ε, και θα περάσουμε στη συζήτηση. Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Συνήθως ε, με καλή η Επιτροπή ΣΕΝΤΕ, η Υποπιτροπή Άμυνα, είναι ενδιαφέρον που με καλέσατε κι εσείς. Είδα ποιε είναι οι αρμοδιότητε τη Επιτροπή σα ε, για να δω τι περιμένετε από μένα αν συζητήσουμε την καταπολέμηση τη πειρατεία στο κέρα τη Αφρική αν δω ε, την περιγραφή των κατοικώντων σας δεν αναφέρονται ούτε η άμυνα ούτε τα στρατιωτικά ζητήματα και είναι λογικό γιατί δεν ε, πρόκειται για επιβολή της νομοθεσίας αλλά πολλά από τα κράτη-μέλη και στις επιχειρήσεις τους ε, υποστηρίζουν την επιβολή του νόμου. Και φυσικά σε πάρα πολλά μέρη όπου έχουμε οργανωμένο έγκλημα έχουμε αστάθεια και τις συνέπειες του οργανωμένου εγκλήματος που επίσης μπορούν να σχετίζονται με τις δράσεις που απαιτούνται από μας να αναλάβουμε. Θα συμφωνήσω με όλους ότι η πειρατεία είναι ένα είδος οργανωμένου εγκλήματος και εμπλεκόμαστε εκεί και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό παράδειγμα που παντρεύετε αυτά τα θέματα και σας ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία να τα συζητήσουμε. Είδα ότι μία από τις ευθύνες σας ε, είναι να δείτε ποιες απειλές υπάρχουν κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και μπορώ να φανταστώ ότι ήδη συμφωνείτε μαζί μου για το πώ η πειρατεία απειλεί τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσετε και πώ το βλέπουμε κι εμεί. Η πειρατεία φυσικά απειλεί τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι από οποιοδήποτε σκάφους, αλλά επίσης απειλεί τη σταθερότητα στην περιοχή με συνέπειες οικονομικές, διπλωματικές, πολιτικές. Είναι δύσκολες οι δράσεις ε, της αντεξής συνεργασίας, υπάρχουν πάρα πολλά project, αλλά η αναπτυξιακή συνεργασία είναι τώρα ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια και δεν υπάρχει ασφάλεια και χωρίς ε, ανάπτυξη, μου είπε ένα συνάδελφος και εγώ συμφωνώ μαζί του. Σίγουρα η πειρατεία προστίθεται στην ανθρωπιστική καταστροφή που έχουμε στη Σομαλία. Δεν είναι μόνο η αιτία, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση εμπλέκεται στην ανθρωπιστική βοήθεια μέσω της ΓΔΕΚΟ. Αλλά και εδώ βλέπουν ότι είναι απαραίτητο να δημιουργήσουν ασφάλεια για τον πληθυσμό πριν να μπορέσουν να είναι αποτελεσματικά τα υπόλοιπα project που τίθενται σε εφαρμογή. Φυσικά αποτελεί και πηγή τρομοκρατικών απειλών έναντι των δυτικών συμφερόντων γενικά και ένας λόγος είναι οι ροές χρημάτων προς την Αλσαμπάμπ που συνδέεται με την Αλκάιντα. Και ένα τμήμα των χρημάτων επίσης ρέπε στο οργανωμένο έγκλημα προς τέτοιους κύκλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν υπάρχουν πολύ καλοί λόγοι για τους οποίους ε, εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και θα ήθελα να τονίσω ότι τα στρατιωτικά δεν είναι τα μόνα μέσα για την καταπολέμηση τη πειρατεία. Εμείς είμαστε μόνο ένα από τα πολλά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με άλλου εταίρου και κρατημέλη. που πιστεύω ότι μπορούμε να πούμε ότι η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι όπω το βλέπω εγώ καθώ έχω εργαστεί και σε άλλους οργανισμού, είναι η καθολική προσέγγιση, όπως την αποκαλούμε τώρα, comprehensive approach, δηλαδή να ομαδοποιούμε όλα τα διάφορα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα κοινό στόχο και η καταπολέμηση της πειρατείας αποτελεί ένα καλό παράδειγμα αυτού. Έχουμε μια στρατηγική πλαισίου με τους γενικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν πάμε ένα βήμα πιο κάτω, ένας από τους στόχους ε, είναι να αντιμετωπιστεί η πειρατεία. Έχουμε ένα σχέδιο δράσης ε, κατά της πειρατεία. Δεν είναι στρατιωτικό σχέδιο αυτό, αλλά αναπτύσσεται υπό την ευθύνη του Διευθύντου με το ε, τμήμα διαχείρισης κρίσεων και σε συντονισμό όχι μόνο με το Συμβούλιο και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, αλλά και με υπηρεσίες της Κομισιόν, όπως η Αναπτυξιακή Συνεργασία και η ΕΚΟ. Μαζί τους ε, διερευνούμε πώς θα φτάσουμε στον τελικό σκοπό, στο τελικό, στην τελική κατάσταση. Η τελική κατάσταση είναι η εξή. Θα πρέπει να αντιμετωπίζει την πειρατεία η περιοχή η ίδια από μόνη της και έχουμε και άλλους στόχους, υποστόχους και είναι λογικό γιατί οι υποστόχοι είναι οι εξής. Όσο υπάρχει πειρατεία πρέπει να καταπολεμάσει τους πειρατές. Αλλά εδώ δεν μιλάμε μόνο για στρατιωτική δράση, αυτό είναι ένα τμήμα. Η δίωξη των πειρατών επίσης ανήκει στην καταπολέμηση της πειρατείας. Πρέπει λοιπόν όλοι αυτοί οι παίκτες να δράσουν στην καταπολέμηση της πειρατείας. Επίσης, Πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες στην περιοχή να αναπτύξουν τις δικές τους ικανότητες έτσι ώστε να μπορέσουν οι ίδιες να καταπολεμήσουν τους πειρατές. Και δεν μιλάμε μόνο για το ναυτικό, μιλάμε και για την ακτοφυλακή. Χρειάζεται να υπάρχουν και δικαστικά συστήματα και όλο το σύστημα επιβολής του νόμου. Επομένως, και εκεί συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν έχει καθόλου στρατιωτική φύση, αλλά είναι μόνο χρήσιμο ε, να κατα... όπως καταπολεμά ο στρατός τους πειρατές της θάλασσα θα είναι αποτελεσματική δράση του μόνο αν συνδυαστεί και με τις υπόλοιπες δράσεις. Και ένας άλλος στόχος είναι πριν το χάρη αν ε, επιτυχώς πολεμήσουμε τους πειρατές, θα πρέπει να δημιουργήσουμε εναλλακτικού τρόπους ζωής για αυτές τις μεγάλες κοινότητες που κερδίζουν πολλά χρήματα μέσω της πειρατείας. Ούτε και αυτό έχει στρατιωτική φύση, αλλά θα πρέπει να γίνει. Και πρέπει να γίνει με μια λογική σειρά. Γι' αυτό το λόγο καθόμαστε γύρω από το τραπέζι με όλους αυτούς τους διαφορετικούς εκπροσώπους, και προσπαθούμε να καθορίσουμε τις δράσεις μας σε μια λογική σειρά. Φυσικά μία από τις άλλες πτυχές είναι ότι πρέπει να συντονιστούμε με όλους τους άλλους διεθνείς εταίρους που επίσης καταπολεμούν την πειρατεία στην ε, ίδια περιοχή. Οργανώσεις όπως το Ηνωμένα Έθνη, αλλά και άλλοι εταίροι όπως Ινδία, η Ιαπωνία, οι Ηνωμένε Πολιτείε και άλλοι που για τα δικά τους συμφέροντα καταπολεμούν την πειρατεία στην ίδια περιοχή και συντονιζόμαστε μαζί τους. Τώρα, ποιο είναι το νομικό μας ε, πλαίσιο. Υποθέτω ότι και αυτό σας ενδιαφέρει. Για μένα ξεκινά με τη βάση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο η κοινή δράση του Συμβουλίου του 2008. Είχαμε και αρκετές τροπήσεις από αυτές. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτή και είναι η δράση του Συμβουλίου συνάδει πλήρως με πολλά άλλα νομοθετήματα διεθνούς και εθνικού δικαίου. με την ε, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, με διάφορα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ, Χρειαζόμαστε κοινοποίηση από την κυβέρνηση τη Ομαλία, το Γενικό Γραμματέα του ΙΕΠ, να μας επιτρέπει να αναλαμβάνουμε δράσεις στα χωρία ύδατα και στα ιστορικά ύδατα και στις παράκτης περιοχές. Έχουμε μια απόφαση της ευρωπαϊκή Ένωσης, του Συμβουλίου, που συμφωνεί με το σχέδιο και με τους κανόνες δέσμευσης που περιγράφουν υπό ποιε συνθήκε εμείς στρατιωτικοί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη βία. Είναι πολύ βασικό αυτό το έγγραφο για μας και πρέπει να μείνουμε αυστηρά μέσα σε αυτά τα όρια, γιατί αν όχι, τότε θα σκηθεί δίωξη στην πατρίδα μας εναντίον μα και έχουμε παραδείγματα αυτού. Κατόπιν έχουμε απόφαση του Συμβουλίου του 2010 που επέτρεψε την επιχείρηση Αταλάντη κατά της πειρατείας ε, να μεταφέρει δεδομένα, να διαβάσει δεδομένα στην Interpol και μέσω της Interpol φυσικά στη Europol. Κατόπιν, συμφωνίες ε, μεταβίμασης, μεταφοράς ε, για την παράδοση των συλληφθέντων πειρατών σε άλλες χώρες, Χέλες και Μαυρίκιο αυτή τη στιγμή. Αυτό καθορίζει το νομικό πλαίσιο για την επιχείρηση Αταλάντη, αλλά κάθε έθνος ε, που συνεισφέρει με στρατό και η πλήρχη κινούνται δυνάμει της εθνικής τους νομοθεσίας. Ε, δεν μπορούν να διευρύνουν την εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μπορεί, παραδείγματος χάρη, να περιοριστεί αυτή η εντολή. Αυτά για το νομικό πλαίσιο. Αν έχετε και άλλες ερωτήσεις, φυσικά είμαι στη διάθεσή σας. Τώρα, για την ίδια την Αταλάντη. Με την ε, UNAFOR, όπως την αποκαλούν. Είναι ο οργανισμός που υλοποιεί την επιχείρηση. Σήμερα αποτελείται από 5 7 σκάφη και 3 ως 5 NPRAs, δηλαδή αεροσκάφη για περιπολίες και αναγνώριση. Και ο προβλέψιμος είναι 8 εκατομμύρια το χρόνο. Τα κράτη-μέλη που δεσμεύουν δυνάμεις βέβαια σηκώνουν και ένα μέρος ε, του άχθους του οικονομικού. Τι κάνουν ακριβώς καταρχήν. Δημιουργούν κατάσταση επαγρύπνησης έχουν ε, τρόπους για ανταλλαγή στρατιωτικών πληροφοριών με άλλους, αλλά και τα πειραίες ε, πίσω ε, στέλνουν πληροφορίε για το που βρίσκονται οι πειρατέ και μέσω από δορυφόρων που βρίσκονται οι πειρατέ είτε στη στην ξηρά. Η ύψιστη προτεραιότητα είναι να διασφαλίσουν την αποστολή του Παγκόσμιου Επιστημιστικού προγράμματο. Αυτή είναι η υψηλότερη προτεραιότητα, η ύψιστη προτεραιότητα στην εντολή για τον επικεφαλή τη αταλάντη. Οι επόμενε προτεραιότητες είναι να διασφαλιστεί οποιαδήποτε άλλη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας και της αποστολή της Αμεζόν, τη αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία, που βοηθά την κυβέρνηση της Σομαλίας ε, να καταστήσει τη χώρα ασφαλή. Κατόπιν, επόμενο καθήκον να αποτρέψει και να καταστήλει την, και να προκαλάβει την πειρατεία και στη θάλασσα και στην ξηρά, στη Σομαλία. Κατόπιν έχει την εντολή να συλλάβει, να να ξελαμβάνει, να κρατά και να μεταφέρει σε νόμιμες αρχές και τονίζεται ότι πρέπει να γίνεται αυτό σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και με το σοβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κατόπιν, μπορούν να συλλεγούν πληροφορίες. Τι είδου πληροφορίες? Αποδεικτικά στοιχεία. Έχουμε εικόνες και βίντεο από τα αεροσκάφη, μπορούν ε, να βγάζουν φωτογραφίες και διαβατήρια με επιδροματικά στοιχεία όταν συλλαμβάνουν και κρατούν τους πειρατές και επίσης μπορούν να δώσουν ε, στοιχεία στην Interpol. Στοιχεία σχετικά με αποδείξεις, αποδεικτικά στοιχεία για τους ε, πειρατές που συλλαμβάνονται. Μέσω της Interpol ε, πάμε στη Europol. Δηλαδή τα στοιχεία αυτά μέσω της Interpol διαβιβάζονται στη Europol. Έτσι μπορούμε να έχουμε και στενότερη συνεργασία με τη Europol. Τώρα, είναι επιτυχής η Αταλάντη. Ναι, μπορούμε να πούμε. Ήταν ιδιαίτερα επιτυχής. Αλλά όχι μόνη τη. Ε, Σα εξήγησα ότι υπάρχει μια συνολική προσέγγιση τη λοιπόν μαζί με όλου του άλλου εταίρου που επίσης καταπολεμούν την πειρατεία. Μπορώ να πω ότι είμαστε ιδιαίτερα επιτυχεί. Είμαστε 100% επιτυχεί στο να διασφαλίσουμε την αποστολή του Παγκόσμιου προγράμματο. Προγράμματος. Τώρα, έχουμε φτάσει στα 212 πλοία που περνούν και σε αποπικίνδυνες περιοχές και έχουμε ένα τόνο ένα εκατομμύριο τόνους, με συγχωρείτε, τροφίμων που περνούν στη Σομαλία και έτσι προστατεύουμε και την υποστηλή της Amazon. Έχουμε αρκετά πλοία μέχρι τώρα και είναι αυτό πολύ σημαντικό γιατί η Amazon βοηθά την κυβέρνηση της Σομαλίας να προσφέρει ασφάλεια στη Σομαλία και ξέρετε ότι το τελευταίο χρόνο μεγάλη επιτυχία το έπραξαν. κάποια νούμερα. Μέλη από 151 μέλη το 2011, τώρα έχουμε 30 το 2012 μέλη πειρατείας. Δεν είχαμε επιτυχείς δράσεις των πειρατών από το Μάιο και χτες Είχαμε πάλι μια πράξη πειρατεία, αλλά αναχαιτίστηκε. Και το Ολλανδικό σκάφος με την Ατελάντη συνέλαβε και κρατά τους πειρατές ε, ενός από τα πλοία που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την επίθεση. Επιτυχία λοιπόν έχει σημειώθει και πριν δύο χρόνια είχαμε 30 πλοία στα χέρια των πειρατών, ενώ τώρα έχουμε, έχουν μειωθεί αυτά στα τέσσερα. Και φυσικά και τέσσερα πολλά είναι. Λοιπόν, να αναφέρω και κάποια στοιχεία από στρατιωτική σκοπιά. Αν θέλουμε να διώξουμε τους πειρατές, στα περισσότερα στήματα του common law, ξέρετε ότι χρειάζεται κανείς μάρτυρα στο δικαστήριο. Για μας ε, αυτό είναι πολύ δαπανηρό και χρονοβόρο. Γιατί ποιοι είναι ε, οι μάρτυρες στα θύματα. Φυσικά οι εταιρείε το πλήρωμα των πλοίων. Που ανεχέτησε την πυρετική δράση, αλλά αν ε, θέλετε να πάνε οι άνθρωποι αυτοί στο δικαστήριο να καταθέσουν, ε, χάνουμε δυναμικός. Ε, ε, βρήκαμε λοιπόν ότι μπορούν να καταθέσουν μέσω βιντεοδιάσκεψης. Ένα άλλο θέμα είναι ότι η Αταλάντη καταπολεμά τα συμπτώματα στη θάλασσα μόνο. Εμείς είμαστε οι, που, πρώτοι συγγνώμη, που παραδεχτήκαμε ότι είναι η ασπιρίνη που δίνεται κατά το πονοκεφάλαιο, αλλά η πραγματική αρρώστια βρίσκεται στην ξηρά. Θα ήταν ε, λάθος να σταματήσει και να παίρνει ασπιρίνη ενώ έχει ακόμη πονοκέφαλο. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τις αιτίε ε, στην ξηρά. Και το κάνουμε και με κάποιους στρατιωτικούς τρόπους. Έχουμε μία αποστολή εκπαίδευσης, εκπαιδευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταρτίζει τις δυνάμεις ασφαλείας στη Σομαλία και τώρα σημειώνει αρκετή επιτυχία μαζί με το Amazon για τη δημιουργία καλύτερων συνθήκων ασφαλείας στο Μαγκαντήσιο και σε όλο το νότο της Σομαλίας τώρα. Έχουμε μία μη στρατιωτική επιχείρηση Ευρωπαϊκή Πολιτική Αμυντική και Ασφάλειας που βοηθά τη δημιουργία ικανοτήτων στις χώρες της περιοχής αλλά και στη Σομαλία, την ακτοφυλακή και ολόκληρο σύστημα κράτους δικαίου. Έτσι λοιπόν εργαζόμαστε και επί άλλων πτυχών, επί της ξηράς αλλά πραγματικά και η ΕΚΟ και η ΔΕΦΚΟ είναι πολύ ενεργές σε πάρα πολλά project στη Σομαλία. Άλλο ένα ζήτημα, και το γνωρίζουμε, είναι το εξή. Εμείς ε, πολεμούμε τους πειρατές στη θάλασσα, αλλά πρέπει να βρούμε τρόπους πώς μπορούμε να βρούμε τους αρχηγούς και να τους αντιμετωπίσουμε. Και το τελευταίο σκέλος δεν είναι στρατιωτικό. Αν βρει κανεί τους αρχηγούς, τότε υπάρχουν δυνατότητες επιβολής του δικαίου, αλλά Επίσης έχουμε τα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπλοκάρουμε παραδείγματος χάρη και τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Υπάρχει μία μικρή σύνδεση με το στρατιωτικό σκέλος, αν παραδείγματο χάρη όπως ε, και κάναμε, καταστρέψουμε κάποιες μηχανές των πειρατών, πρέπει να αγοράσουν καινούργιε. Αν ε, ξέρουμε από πού τις αγοράζουν, μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις ε, χρηματοοικονομικές ροές. Αλλά πρέπει να καταστρέψουμε αρκετέ μηχανές και να ενημερώσουμε άλλους ότι το πράξαμε. Γιατί το υπόλοιπο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες. Κάτι ακόμη. Καταλαβαίνουμε, θα θέλαμε, αλλά κατανοώ και την Europol να έχουμε στενότερη συνεργασία με την Ευρωπόλ. Νομίζω ότι θα ήταν καλό αν είχαμε και ανταλλαγή πληροφοριών μαζί της. Να στέλνουμε αποδεικτικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσει, αλλά πολλές φορές όσοι δεν μπορούν να δώσουν λεπτομερείς πληροφορίες ε, για άτομα, αν τους δίνουμε εμείς πληροφορίες ότι συλλάβουμε τα άτομα αυτά και έχουμε ονόματα και αποδεκτικά στοιχεία, θα μπορούσαν να μας πούν τι να κάνουμε. Έτσι ώστε να μην ε, αφήσουμε κατά λάθο, να μην απελευθερώσουμε κατά λάθο κάποιου που τελικά θα αποδειχτούν να είναι αρχηγοί των πειρατών. Αυτά μπορεί να είναι θέματα που μπορεί να θέλετε να συζητήσετε και νομίζω ότι μπορώ να κλείσω εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ αντιστράτηγε. Πράγματι, έχουμε ισχυρή αστυνομική και δικαστική παρουσία, αλλά και από μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Πάντως, εσείς είσαστε ο πρώτος στρατιωτικός που μας έρχεται. Ταιριάζουν όμως όσα μας είπατε πολύ καλά στα καθήκοντα της Επιτροπής μας. Αναφερθήκατε λοιπόν στην ανθρωπιστική κρίση στη Σομαλία, πολύ σημαντικά. Και έχουμε βέβαια και τη συνεργασία με τη Europol. Από τη Europol είναι ο κύριος Κώστερ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να έρθω εδώ. Θα περιγράψω κάπως γρήγορα το πώς δουλεύουμε εμείς στην οργάνωσή μας. Ξέρετε ότι δίνουμε επιχειρησιακή στήριξη στις αρχές που ασχολούνται με έρευνες εγκλημάτων. Αυτό είναι λοιπόν το νομικό μας πλαίσιο. Δεν έχουμε εκτελεστικές δραστηριότητε. Κάνουμε την ανάλυση μας και στηρίζουμε τις επιχειρήσεις των κρατών μελών. Έχουμε 200 αναλυτές οι οποίοι δουλεύουν καθημερινά πάνω σε διαφόρους φακέλους. Από το Μέο του 2012 Έχουμε έναν για την, ε, τη δράση κατά της τρομοκρατίας. Έχουμε και διάφορα σημεία focal points. Τι ακριβώς κάνουμε τώρα στη Europol. Από το 2010 ανοίξαμε ε, τον φάκελο για την πειρατεία και κάνουμε διάφορους ελέγχους με συλλογή στοιχείων σε καθημερινή βάση και σε συνεργασία με άλλα focal points. Αναλύουμε τις πληροφορίες λοιπόν που έχουμε σχετικά με το θέμα αυτό. Ό,τι πληροφορίες σχετικές έχουμε στη Europol. λοιπόν υπάρχει ένα θέμα ξεπλήματος χρήματος που συνδέεται με την πειρατεία, εμείς θα αρχίσουμε να ψάχνουμε και στο focal point για το ξέπλυμα χρήματος. Σήμερα το focal point για την πειρατεία έχει να κάνει με 35.000 μονάδες. Πρόκειται για ονόματα, πρόκειται για αριθμούς τηλεφώνου, ε, επικοινωνίες, αλλά μπορεί να είναι DNA, μπορεί να είναι και δαχτυλικά ε, αποτυπώματα. Με 60.000 links ανάμεσα στις μονάδες αυτές. Όλα είναι προς έρευνα. Μετά περνάμε στην σε βάθος ανάλυση, βέβαια λιγότερον. Το δεύτερο εξάμεινο του 2010 είχαμε 36.000 υποθέσεις που ερευνήσαμε που είχαν να κάνουν με υποτυπώματα DNA. 12 ε, χώρες ε, μέλη συνδέονται με τα focal points αλλά και οι Ηνωμένε Πολιτείε, ε, σχετικές ερευνητικές οργανώσεις, δύο ερευνητικά Ινστιτούτα, Eurojust και η Interpol. Έχουμε επίσης την Joint Investigation Team Operation Nemesis. Την πρωτοβουλία της Ολλανδικής Συγγελίας υπάρχει μια μεικτή ομάδα που ονομάζεται Nemesis και η οποία ξεκίνησε από το 2012 και στηρίζεται βέβαια από εμά από την Europol και την Eurojust. Αποτελείται από την Ολλανδία και τη Γερμανία και ουσιαστικά φιλοξενείται από την Europol. Είναι η πρώτη φορά ουσιαστικά που ένα JIT ε, φιλοξενείται στην Europol. Δηλαδή για πρώτη φορά ανακριτές ε, από τη Γερμανία και την Ολλανδία κάθονται μαζί με μια ομάδα αναλυτών της Europol μέσα στην Europol. Αυτό από μόνο του έχει τεράστια αξία, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει μόνιμη σχέση ανάμεσα στην ανάλυση και αυτούς που δουλεύουν στην JIT. Θέλω να σας ενημερώσω για τα προκαταρτικά μας αποτελέσματα που φαίνεται ότι είναι πολύ βελτιωμένα. Ο στόχος της Joint Investigation Team, αυτής της JIT που λέγαμε, της μικτής δηλαδή ερευνητικής ομάδας, είναι η οργάνωση, τα δημοσιονομικά, Όσοι ασχολούνται με την ε, πειρατεία είναι βέβαια γνωστοί αυτοί οι άνθρωποι ανήκουν στην λίτ ε, συνήθως την κοινωνική και την οικονομική της ε, χώρας και προστατεύονται από υψηλή διπλωματική προστασία. Ο εντοπισμός λοιπόν των ατόμων μέσα σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ασταθές, χωρίς κεντρική κυβέρνηση, ή συγκεκριμένα αρχεία πολιτών, καταλαβαίνετε ότι αποτελεί ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Πολύ συχνά ε, τους ανθρώπους τους γνωρίζει κανείς μόνο με ένα ψευδόνυμο ή το μικρό του όνομα και όχι με το επίθετο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το DNA, τα δακτυλικά αποτυπώματα, είναι ο μόνος τρόπος που έχουμε για να εντοπίζουμε τους δράστες. Τώρα τα χρήματα. Είναι και αυτό μια δύσκολη επιχείρηση. Με τα χρήματα δεν γίνεται. Πηγαίνουν μέσα σε σάκους, σε ένα συγκεκριμένο σημείο που τα παίρνουν οι δράστες και μεταφέρονται μέσα από συστήματα εντελώ άτυπα. Σπάνια εμφανίζονται τραπεζικοί, οργα... τραπεζικοί λογαριασμοί. Και τα ποσά αυτά μετά επενδύονται είτε για αγορά γης, είτε σε εγκληματικέ ε, δραστηριότητες, ναρκωτικά για παράδειγμα. Εμείς βασιζόμαστε κυρίως σε στοιχεία που έχουμε από τις επικοινωνίες για να αναλύσουμε τα δεδομένα που έχουμε. Βασιζόμαστε δηλαδή στις πληροφορίες που μας φτάνουν από τους διαπραγματευτές. Η επικοινωνία έτσι μας βοηθάει να ε, ξαναβρούμε την άκρη με τα δίκτυα. Έχουμε να κάνουμε το οργανωμένο έγκλημα, δεν έχουμε να κάνουμε τρομοκρατία. Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι αναμειγνύονται τρομοκρατικές οργανώσεις στην πειρατεία στη θάλασσα. Είναι πολύ ασφαλές, μπορούμε δηλαδή κάλλιστα να πούμε ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα και τις εγκληματικέ οργανώσεις που η ΑΣΟΠΑΠ είναι μια ε, οργάνωση εγκληματική και τελικά φτάνουμε να πιστεύουμε ότι πληρώνεται και κάτι σαν επαναστατικός φόρος. Αλλά αυτός είναι ο λόγος που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα στο focal point για την πειρατεία το θέμα αυτό. Και να ξέρετε ότι στην Αφρική δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με αυτό. Έχουμε και την Ιεμένη, έχουμε και την ε, Αλκαΐδα. Που σε καθημερινή βάση είναι σε επαφή μεταξύ τους, είτε για θέματα κατάρτισης, είτε άλλα. εκπαίδευση δηλαδή των μαχητών τους κλπ. Κάτω το παρελθόν, αυτό που προηγήθηκε του Βασεμπάκ, αντιμετώπιζε ως ε, Ισλαμιστικές οργανώσεις αυτές. Μετά όμως στη συνέχεια και μετά τον πόλεμο άλλαξε η στάση του Ασεμπάπ στον τομέα αυτών. Τι άλλες προκλήσεις έχουμε. Η ανταλλαγή πληροφοριών λοιπόν είναι το βασικό για, την, ε, για το συντονισμό. Εμπλέκονται εδώ και στρατιωτικοί παράγοντες. Αυτό που απασχολεί πάντως στη Europol είναι να έχει περισσότερες πληροφορίες από την Ατλάντα. με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τη συμμετοχή ειδικών από την στρατιωτική πλευρά, αλλά και από τη δικιά μας την πλευρά και γι' αυτό είμαι πολύ ικανοποιημένο ε, από τη συνεργασία που έχουμε με την UNIFOR. Αλλά το είπατε κι εσείς λίγο πολύ, ότι χρειαζόμαστε απευθείας επαφή ανάμεσα σε μία αποστολή STIP και τις δικές μας ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Αν δεν είναι στρατιωτικές αποστολές αυτές, τότε αυτό πρέπει να γίνεται μέσω μιας χώρας. Δεν μπορούμε να έχουμε ανταλλαγή απόψεων βάσει του νομικού μας πλαισίου με αποστολές CSDP. Θέλουμε να αλλάξουμε φυσικά την κατάσταση αυτή, αλλά είμαστε αστυνομικοί και από μεριά έχουμε τους στρατιωτικούς που είναι γνωστοί για την πραγματιστική τους προσέγγιση. Και εμείς αυτή την πραγματιστική προσέγγιση θέλουμε πάντοτε. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι να βοηθήσουμε στην Αταλάντα όσο γίνεται περισσότερο και με όσο γίνεται πιο ήπιο τρόπο. Αν δεν μπορούμε να ανταλλάσσουμε απευθείας πληροφορίες με την ΓΕΝΑΦΟΡ, τότε Έχουμε και την υπηρεσία εξωτερικής ε, δράσης. Αλλά στο μεταξύ έχουμε καθημερινή επαφή και ανταλλαγή πληροφοριών με την UNAFA. Ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ πολύ. Ερωτήσεις έχουμε από την κυρία Μόρφα και τον κύριο Νιούτον Ντάν. Κυρία Μόρφα, ευχαριστώ πολύ και τους δύο μιλητές όπως σωστά είπε ο Πρόεδρος, έχουμε συνθήσει στη ΣΕΝΤΕ να καλούμε ανώτερους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων που εμείς ασχολούμεθα με θέματα εγκλήματος και ε, ως επιτοπλίστων συνεργαζόμεθα και συνομιλούμε την αστυνομία και όχι τις ενόπλες δυνάμεις. Η ερώτησή μου τώρα. σε ποιο βαθμό τηρείται η αρχή της ε, αναλογικότητας ε, και της αναγκαιότητας ε, σε ποιο βαθμό ισχύουν αυτές οι αρχές στις ένοπλες δυνάμεις σε σχέση με την αστυνομία γιατί δεν ξέρω έχετε καθόλου στατιστικά στοιχεία φαντάζομαι πως διενεργούνται οι επιχειρήσεις αυτές Πολλές φορές χρησιμοποιείτε όπλα. Ε, τι κανονισμοί ισχύουν για σας, γιατί όταν μιλάμε για το έγκλημα γενικά και τις διοκτικές αρχές, ε, τις αστυνομικέ αρχές στην Ευρώπη, εκεί είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Εσείς τι κανονισμούς έχετε και τι στατιστικά στοιχεία υπάρχουν για απώλειες ανθρώπινων ζώων και τραυματισμούς των δραστών στα πλαίσια μιας στρατιωτικής επιχείρησης. Δεύτερη ερώτηση που έχει σχέση με την πρώτη. Θα ήθελα να μου πούν και οι δύο ομιλητές να μα πούν περισσότερα πράγματα για το εμπειρατεία σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα, ως μορφή οργανωμένου εγκλήματος. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν ομοιότητες και με άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος, θέσεις εξουσίας κλπ. Αλλά οι δράστες που βλέπετε εσείς ως στρατιωτικοί στις στρατιωτικές επιχειρήσεις ποιοι είναι. Μήπως είναι οι φτωχότεροι, μήπως είναι πιο ευάλωτοι από αυτά τα κυκλώματα. Δηλαδή φαντάζομαι ας πούμε σε κοινωνικό ή εγκληματολογικό ή κοινωνιολογικό επίπεδο μοιάζουν λίγο με τα βαποράκια, είναι κάτι ανάλογο στα πλαίσια της διακίνησης ναρκωτικών. Δεν είναι δηλαδή ψηλά ιστάμενοι δεν είναι αυτοί που βγάζουν τα πολλά χρήματα. Δεν ξέρω, υποθέσεις κάνω, σε ποιο βαθμό ε, είναι αυτοί οι άνθρωποι που είναι οι πιο ευάλωτοι, παρόλο που διαπράττουν ε, επικίνδυνα προφανώς ε, εγκλήματα, δεν αμφιβάλλω εδώ καθόλου, αλλά πείτε μου έχω δίκιο στις υποθέσεις μου. Και πώς αντιμετωπίζονται οι εγκληματίες αυτοί από την Ευρώπη και τις ευρωπαϊκές διοκτικές αρχές και τις αρχές επιβολής του νόμου. Ο κύριος Νιούτον Τζαν, Νταν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, μ' αρέσει που βλέπω στρατιωτική στολή στην Επιτροπή γιατί συνήθως ε, είναι ανιάρα τα ρούχα που φοράμε, εκτό αν φοράνε ωραία πράγματα οι κυρίες. Αυτή τώρα τι είναι εθνική στρατιωτική ε, στολή ή ευρωπαϊκή. Γιατί είστε στην ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, οπότε μπορεί να είναι η ευρωπαικη γιατι ειστε στην ευρωπαικη υπηρεσια εξωτερικη δραση οποτε μπορει να ειναι η στολη σα ευρωπαϊκή, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, άλλες ερωτήσεις η ε, πειρατεία γίνεται και στην Ιγυρία από την άλλη μεριά. Εκεί καθόλου τι γίνεται, έχει αναλάβει κάποιος άλλος οργανισμός εντελώς διαφορετικός. Επίσης, είπατε κάτι που με έκανε να ορτσώσω τα αυτιά μου. Είπατε ότι υπάρχουν διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρώπη, αυτή από τη Σομαλία. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Έχετε και άλλες πληροφορίες, λοιπόν, υπάρχουν συμμορίες στην Ευρώπη που οργανώνουν τους Σομαλούς. Τι διασυνδέσεις υπάρχουν, τι κάνουν ε, αυτοί από κοινού. Ευχαριστώ κύριο Στάσνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ στρατηγέ μου. Ευχαριστώ και τον κύριο Κώστερς για την, ε, τις εξαιρετικές, ευχαριστώ και τους δύο μιλητές, εξαιρετικά αυτά που μας είπατε. Εγώ βλέπω στρατιωτικού στην Επιτροπή ΣΕΝΤΕ και σας συγχαίρω για την επιχείρηση Αταλάντα που έχει ορατότητα, είναι διακριτός ο ρόλος της και έχει σχέση με πολλά από αυτά που κάνουμε κι εμείς. Ξέρουμε τις επιχειρήσεις αυτές και βέβαια αν έχουν επιχείρηση, δρούν πολλαπλασιαστικά. Χαίρομαι που η Αταλάντη στην Ανατολική Ακτή ε, παίζει ρόλο και για την ε, δημιουργία σταθερότερης κυβέρνησης Σομαλία. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που είπαν και προηγούμενοι συνάδελφοι. Μπορεί να υπάρξει μετατόπιση προς Ανατολάς. Βλέπε Μαλή. Υπάρχει εδώ συνεργασία λόγω κοινών συμφερόντων. Πολλοί συμμετέχουν στις μεταφορές λαθ εχθρέων προϊόντων, μπορεί να είναι όργανα ανθρώπινα ή προϊόντα. Και τέλος, οι τελευταίες αγορές, οι τελικές αγορές είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην, ε, στις ΕΠΑ και συνεργασία υπάρχει, γιατί οι τελικές αγορές μπορεί να είναι σε πολλά μέρη του κόσμου. Η τελευταία είδαμε πειρατεία στην Ανατολική Αφρική, στις Ανατολικές Ακτές. Αυτό πώς αξιολογείται. Είναι νέα τάση ή είναι μεμονωμένο συμβάν. Αν ισχύει το πρώτο είναι πολύ ανησυχητικό. Ε, και οι στρατιωτικοί μας τι βλέπουν ως επιλογές ε, για την αντίδρασή μας. Είναι αυτό ε, ένας πονοκέφαλος. Τέλος για τα χρήματα Χαίρομαι που αναφέρθηκε, γιατί αναρωτιόμουν πού τα βρίσκουν τα χρήματα. Συνήθως είναι μετρητά. Αλλά και γι' αυτό πώς παρακολουθείτε το ίχνος του χρήματος. Βλέπω ότι γίνεται, γιατί βλέπετε να ανθούν επιχειρήσεις, να υπάρχει ευημερία. Οπότε ε, εκεί ε, μπορείτε να ε, δείτε ποιοι είναι αυτή, που δεν είναι εκατοντάδες ή χιλιάδες, μπορεί να είναι κάποιες ε, δεκάδες άνθρωποι. Και όταν εντοπίσουμε την ε, δραστηριότητα σταματούν ή μπορεί να βρουν άλλες περιοχές, άλλα πεδία δράσης. Να, ο, ίσως αυτό να είναι ένα παράδειγμα η μετατόπιση στην, στην Ανατολική Αφρική. Η κυρία Βάιλερ. Δύο σύντομες παρατηρήσεις. Ίσως είμαι λίγο παλαιομοδίτησα, αλλά διαβάζοντας ε, τις εφημερίδες ε, και ακούγοντας τα ΜΜΕ, βλέπουμε ότι η μάχη κατά της πειρατείας συνδέεται αναπόφευκτα με την καταπολέμηση της ε, φτώχειας. Και αν δεν γίνει κάτι σε αυτό το μέτωπο, κατά πάσα πιθανότητα θα εξακολουθήσουμε να έχουμε τέτοια αποτελέσματα γιατί υπάρχει μια γκρίζα ζώνη και σε νομικό επίπεδο. Θυμάστε στη Γερμανία, στο Αμβούργο που έγινε μια δίκη ε, κατά των δραστών και είδαμε πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά με τη βοήθεια εσωτερικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Πιο καλά λοιπόν θα ήταν να αρχίσουμε μάχη κατά της φτώχειας εκεί. Αυτό είναι ένα που ήθελα να πω. Δεύτερον, θα ήθελα μια εκτίμηση με βάση την πείρα σας. Ε, ο σκοπός της Επιτροπής κρίμηνε να δει αν μπορούμε να ε, εισάγουμε, τον εισαγάγουμε τον θεσμό του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα με παρόμοιο τρόπο όπως λειτουργεί αυτό στη ΣΥΠΑ. Εσείς πώς το βλέπετε. Η δράση σας ε, συνοδεύονται από την απαραίτητη υποστήριξη ή πιστεύετε ότι πρέπει να, έχουμε, ε, να θεσπίσουμε το, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ευχαριστώ. Κάποιες ερωτήσεις και από μένα. Κύριε Αντιστράτηγε, είπατε ότι ο κυβερνήτης του σκάφους είναι, υπόκειται στο δίκαιο που διέπει το σκάφος και αν είναι με σημαία ευκαιρίας, τι γίνεται. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πολλά από αυτά τα σκάφη είναι ιδιοκτησία ευρωπαϊκών ή αμερικανικών ε, ναυτιλιακών εταιριών ή ε, εταιριών από άλλα μέρη του κόσμου. Αλλά ένα μεγάλο ποσοστό είναι του Παναμά, της Λιβερίας και άλλες τέτοιες χώρες. Και τότε, τι ευθύνη έχουν αυτές οι εταιρείε που βάζουν τα σκάφη κάτω από τη δικαιοδοσία του Παναμά, αλλά μετά δεν περιμένουν βέβαια από το ναυτικό του Παναμά να πάει να τα σώσει στο κέρας της Αφρικής. Και μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό των σημείων ευκαιρίας από το διεθνές δίκαιο. Δεύτερον, διάβασα για την πόντιση επικίνδυνων ε, ε, ουσιών και προϊόντων στα ύδατα της Σομαλίας. Από τρίτους. Ακόμα και πυρηνικά απόβλητα άκουσα ότι ποντίζονται εκεί. Είναι αυτό μέρος της εντολής σας. Και αν, θα, αν είναι ή αν ήταν αυτό μέρος της εντολής σας, θα βοηθούσε στην καταπολέμηση του εγκλήματος εκεί, αν θα μπορούσε δηλαδή να ισχύσει το κράτος δικαίου ε, εκεί, στα τα αυτά. Θα μπορούσε δηλαδή από εκεί να ε, ε, εφαρμοστεί και το κράτος δικαίου σε, άλλες, σε άλλους τομείς. Επίσης, ε, αυτά τα ε, σκάφη, τα μη επανδρομένα ε, που παρακολουθούν, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ή είναι μόνο για την ξηρά σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Τον κύριο Κώστερς, ξέρω ότι υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών αλλά διαβαθμισμένων σε μεγάλο βαθμό. Τώρα, για την εφαρμογή του TFTP, όταν ε, εγκρίναμε τη δεύτερη συμφωνία TFTP με τη ΣΥΠΑ, ε, πρέπει κυρίως να δράσουμε στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά και σοβαρό διακρατικό, το σοβαρό διακρατικό έγκλημα. Και πολλές φορές η Europol δίνει άμεσα απευθείας πληροφορίες στη ΣΥΠΑ. Και εις αντάλλαγμα τι παίρνουμε. Παίρνουμε κάποια ε, χρήσιμα στοιχεία. Δεν θέλω ε, πληροφόρηση ενημερωμένη, αλλά ε, αξιοποιείτε την πληροφόρηση που σας δίνουν για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, εκτός από την πειρατεία. Και ένα σχόλιο τέλος Η Europol δεν έχει εκτελεστικές εξουσίες και είναι λίγο περιορισμένη σε σχέση με τις πληροφορίες που θα δώσετε, ας πούμε, στη δικαστική εξουσία και όχι στις, επιχειρήσεις του στρατού. Τέλος, ε... ίσως αυτό θα πρέπει να, γίνει ένα ερώτημα, να είναι ένα ερώτημα που θα γίνει στο μέλλον. Τέλος, ο κύριος Βανόλς και ο κύριος Κώστερς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για αυτές τις ενδιαφέρουσες ε, ερωτήσεις. Σε σχέση με τους κανονισμούς για τη στρατιωτική χρήση, συγκρίνεται με το τι ισχύει για την αστυνομία. Γιατί η ρύθμιση είναι πάρα πολύ αυστηρή, το πότε δηλαδή θα χρησιμοποιηθεί η βία ισχύει. Και αυτό ε, ισχύει για κάθε αποστολή. Υπάρχει και εντολή από το Συμβούλιο και στη δική μας περίπτωση αλλά και σε εθνικό επίπεδο ο εθνικός διοικητής λαμβάνει και εθνικές οδηγίες αν υπάρχουν περιορισμοί στους ευρωπαϊκούς κανόνες. Και οι κανόνες της δέσμευσης, ε, της παρέμβασης θα πρέπει πάντοτε να συνάδουν με την εντολή. Επομένως ε, και ο διοικητής και όλα τα πλοία και τα αεροσκάφη στην Αταλάντη έχουν ε, ένα σύνολο κανόνων ε, για τις παρεμβάσεις που περιγράφουν ότι σε ποιες συνθήκες μπορούν να χρησιμοποιήσουν όπλα ή γενικά ισχύ. Αν βγει κανείς εκτός της εντολής, τότε θα ασκηθεί δίωξη εναντίον του. Και αν ε, υπάρχουν ε, τραυματίες, ε, είτε από την πλευρά των πυρετών είτε από τη δική μας, θα υπάρξουν έρευνες που θα γίνουν από τις αρχές επιβολής του νόμου για το περιστατικό αυτό. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Μπορεί να υπάρξει και δικαστήριο πίσω στη χώρα για να ερευνήσει αν έχουν γίνει σεβαστοί κανόνες. Τώρα, αν έχω στατιστικά στοιχεία αυτή τη στιγμή, όχι δεν έχω. Αν ψάχναμε, σίγουρα θα μπορούσαμε να βρούμε κάποια νούμερα. Ναι, υπάρχουν και πειρατές ε, που σκοτώθηκαν πάνω στην επιχείρηση, όμως αυτό το εξετάζουν οι αρμόδιοι επιβολείς του νόμου. Η το στρατιωτικό σκέλος έχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την ισχύ και βέβαια ε, εξαρτάται τη ισχύ από στους, μάλλον στους εθνικούς κανόνες. Κάποιοι θα πρέπει να έρθουν άμεσα σε επαφή με τους ε, αξιωματικούς των διοικητικών αρχών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν αυτοί οι αξιωματικοί επί τους σκάφους. Έτσι λοιπόν σε πολλές περιπτώσεις είναι εύκολο, γιατί και αυτοί θα συμμετέχουν στην συλλογή των αποδεκτικών στοιχείων. Όμω, ε, σε κάθε πλοίο υπάρχουν αυστηροί κανόνες για το πώς συλλεγόνται αυτά τα αποδεκτικά στοιχεία. Αυτό γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της Interpol. Χρησιμοποιούμε λοιπόν ε, το ίδιο ομορφότυπο γιατί θα πρέπει να συλλέγονται οι αποδείξεις με ένα σωστό τρόπο, διαφορετικά είναι άχρηστο στο δικαστήριο. Και τολμώ να πω ότι οι εμπειρίες που έχουμε τώρα είναι ότι οι αποδείξεις, τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από την Ελλάδα και έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλές δικαστικές ε, υποθέσεις. Έχουμε φτάσει νομίζω σήμερα στην δίωξη πυρετών. Δεν έχω τον ακριβή αριθμό όσων έχουν φυλακιστεί. Αυτοί έχουν ε, δικαστεί βάσει αποδεικτικών στοιχείων που συλλέχθησαν από την Αταλάντη. Επομένω, γι' αυτό για μένα είναι απόδειξη ότι γίνεται με σωστό τρόπο η συλλογή των στοιχείων, διαφορετικά θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί. Αυτά για τις πρώτες δύο ερωτήσεις σας. Κατόπιν, ε, πειρατές στη θάλασσα. Θα τους συνέκρινα με τους βαρόνους των ναρκωτικών και τους εμπόρους ναρκωτικών. Κάποιοι είναι πρώην ε, αλείς, κάποιοι είναι απλώς, ε, κάποιοι που αναζητούν την περιπέτεια και έρχονται από και θέλουν να κερδίσουν πολλά χρήματα. η επικεφαλής ε, των κλάν συνήθως σε αυτούς δεν αρέσει καθόλου ότι οι νέοι μπαίνουν στην πειρατεία για να κερδίσουν περισσότερο από ό,τι θα κερδίζαν ήταν απλώς αλής. Συχνά ακούω ότι ένας από τους λόγους που έλκονται από την πειρατεία είναι λόγω της ανέχειας. Θα συμφωνούσα αν μπαίναμε σε αυτήν την ερώτηση ότι ναι, πρέπει να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια. Αλλά στην εντολή μας λέμε ότι πρέπει να παρακολουθούμε και την αλία γιατί υπήρξαν καταγγελίες από την σομαλική πλευρά επειδή υπάρχει, είπαν ότι υπάρχει πειρατεία, γιατί υπάρχουν πολύ πιο εξυγχρονισμένα σκάφη ευρωπαϊκά που αλλιεύουν στην περιοχή και υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Όμως δεν υπάρχει παρανομή αλλιέ. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει ανέχεια. Ο λόγος όμως που υπάρχει πειρατεία είναι επειδή μπορούν να κερδίσουν άνθρωποι αυτοί περισσότερα χρήματα. Και κατόπιν, ε, αν δούμε το οργανωμένο έγκλημα, γενικά έχουμε άλλη ορολογία. Αλλά αυτό που κάνουμε και νομίζω το ίδιο κάνει και η Ευρωπόλ. Προσπαθούμε να δούμε ποιο είναι ο κύριο λόγο που έχουμε αυτό το οργανωμένο έγκλημα. Και για εμά, όταν εξετάζουμε την πειρατεία, πρέπει να δούμε ποιο είναι ο κύριο λόγο ύπαρξη τη πειρατεία απάντηση είναι ότι αποτελεί καλή επιχείρηση για τους αρχηγούς που επενδύουν σε αυτή. Και είναι τώρα το κέντρο της βαρύτητας λοιπόν. Το επίκεντρο της βαρύτητας είναι αυτή η αρχηγή. Και γιατί συνεχίζουν αυτοί να επενδύουν στην πειρατεία και να πληρώνουν τους στόχους ομαλούς που δεν κερδίζουν και ιδιαίτερα, αλλά τουλάχιστον κερδίζουν κάτι περισσότερο από ότι να κάνουν οποιαδήποτε άλλη δουλειά στη Σομαλία. επειδή το κόστος, η σχέση κόστος-οφέλους ε, εξακολουθεί να είναι καλή για τους αρχηγούς. Έτσι λοιπόν, ε, αν το όφελος υπερβαίνει πολύ το κόστος, τουλάχιστον πρέπει να αυξήσουμε το κόστος και το κίνδυνο και πρέπει επίσης ε, να εργαστούμε για να μειώνονται τα λίτρα. Αυτό βέβαια είναι και αρμοδίο της εταιρείας που πληρώσει τα λίτρα για να πάρει πίσω το πλήρωμα και το φορτίο. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας, ε, για τη στολή, μου άρεσε. Γιατί και είστε Βρετανός. Αλλά, ξέρετε, δεν έχουμε στολές ε, του ΝΑΤΟ, δεν έχουμε ούτε στολές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί κάθε έθνος λαμβάνει απόφαση για τη χρήση των δικών του στρατιωτικών δυνατοτήτων. Εγώ λοιπόν είμαι Ολλανδός και είμαι αποσπασμένος ειδικός απεσταλμένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί και σε αυτά τα προβλήματα που προσπαθούμε να επιλύσουμε διακυβεύεται και το εθνικό συμφέρον. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Κατόπιν πήρατε ε, στην Ιγυρία. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και εγκληματίε εκεί, αλλά όπω τρει σκοπιά δεν βλέπω κάποιο σύνδεσμο, αλλά πρέπει να το παρακολουθήσουμε στενά αυτό το θέμα, γιατί μπορεί να απειλεί και το δικό μα συμφέρον. Κατά Κατόπιν, σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δώσω κάποια περισσότερα στοιχεία. Το νούμερο που έχουμε δείχνουν ότι πολλά από τα χρήματα παραμένουν και στην περιοχή. Αλλά Υπάρχει προσδοκία και υπάρχουν και αποδείξεις ότι κάποια από τα χρήματα ρέουν και εκτός της ευρύτερης περιοχής και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πλατεία είναι μια νέα τάση. Όχι. Είναι <laughs> πολύ μεγάλη ηλικία, χιλιάδων χρόνων. Είχαμε και πρόβλημα στα στενά της Μαλάκας, έτσι λοιπόν είχαμε κάποια διδάγματα από εκεί, πώς το έλυσαν το θέμα εκεί. Και φυσικά πρέπει να πολεμήσει κανείς τη θάλασσα, αλλά πρέπει να επιλύσει το πρόβλημα στην ψηρά. Τώρα πώς ε, παίρνουν τα χρήματα, ο κύριος ήδη απάντησε εν μέρη. Δεν ε, είναι εύκολο να τα παρακολουθήσουμε, είναι μετρητά αλλά αν αγοράσει κανεί τα πράγματα που χρειάζεται στι μεγάλες εταιρείε, μπορεί να προσπαθήσει να εντοπίσει και να βρει αυτέ τι ε, χρηματοοικονομικές ζωέ Πολύ δύσκολο, δεν ε, είναι δικό μου καθήκον και καλή τύχη στην Γεροπόλ και στην Ιντερπόλ και σε όποιον άλλον τα διερευνά αυτά. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Απάντησα εν μέρη. Η φτώχεια είναι ένα πρόβλημα, αλλά θέλω να πω δύο πράγματα. Το ένα είναι επανάληψη αυτού που είπα, δηλαδή ότι στο βαθμό που οποιοδήποτε μπορεί να κερδίσει περισσότερα από αυτή τη δουλειά, από ότι ε, μέσα από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη δραστηριότητα, ε, πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να βγάλουν περισσότερα χρήματα και θα το κάνουν αυτό. Ένα άλλο σημαντικό επιχείρημα και μπορείτε να ρωτήσετε και την Ανάπτυξη και την ΕΚΟ ποιος ε, του στηρίζει εκεί. Γιατί βλέπουμε ότι επενδύουν πολλά χρήματα, ε, επενδύονται πολλά χρήματα σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, στην καταπολέμηση της φτώχειας και παρόλα αυτά όμως συνεχίζουν. Αν δεν υπάρχει ασφάλεια, οι δραστηριότητες οι παράνομες συνεχίζονται. Πρέπει να βοηθήσουμε λοιπόν την σομαλική κυβέρνηση και σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο να δημιουργήσει κλίμα ασφάλειας. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει και αυτό κάνουμε. Η καταπολέμηση της πειρατείας είναι ένας τομέα. Η εκπαίδευση της ακτοφυλακής, των σωμάτων ασφαλείας, των δυνάμεων ασφαλείας είναι ένα άλλο επίπεδο. Θα πρέπει όλο το σύστημα της επιβολής του νόμου να ε, βελτιωθεί ε, φυλακές για να παραδίδονται και εκεί οι πειρατές γιατί θα πρέπει να τηρούνται τα πρότυπα που έχουμε θέσει. Η καταπολέμηση της φτώχειας είναι λοιπόν ένας ε, τομέας γιατί ε, είναι ένας τομέας όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούμε να συνεργαστούμε και με όλους τους άλλους που πρέπει όλοι να κάνουν τη δουλειά τους για να επιληθεί ριζικά το πρόβλημα. Κύριε Πρόεδρε, με ρωτήσατε κάτι για τις σημαίες ευκαιρίας. Είναι μια δυσκολία αυτή, βεβαίως. Έχουμε πολλά εμπορικά σκάφη, τα οποία είναι ιδιοκτησία μιας εταιρείας και τα πληρώματα μπορεί να είναι από 5 ή 6 διαφορετικές εθνικότητες ποια είναι η ευθύνη των εταιριών. Έχουμε βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης στην Αταλάντη, ε, δίδουμε σε όλες τις εταιρείες αυτές τις πρακτικές και θέλουμε να τις στηρούν. Ποιες είναι, πώς θα διασφαλίσετε καλύτερα το σκάφος, τον εαυτό σας, πώς θα τηρήσετε συγκεκριμένες διαδρομές και να μην πάτε σε επικίνδυνα νερά τα οποία ε, κατέχονται από πειρατές θα πρέπει να υπάρχουν συστήματα πάνω στο σκάφος ούτως ώστε τα πληρώματα να προστατεύονται, να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια από τους πειρατές και να μπορούμε να εντοπίζουμε τους πειρατές χωρίς ζημία στα πληρώματα. Αυτά όλα είναι ευθύνη των ε, ιδιοκτητριών εταιριών. Έχουμε όμως και περιπτώσεις όπου οι ασφαλιστικές εταιρείες ε, δημιουργούν δυσκολίες αν οι εταιρείες δεν ακολουθήσουν αυτές τις βέλτιστες πρακτικές ε, διαχείρισης. Αυξάνουν τα ασφάλιστρα κλπ. Και όλο αυτό το κλίμα νομίζω ότι βοηθάει στην καταπολέμηση της πειρατείας. Τώρα για την δίωξη. Α, κάτι άλλο για τις πλειοκτήτριες εταιρείες ως επιτοπλίστων πρέπει να καταβάλουν εκείνες τα λίτρα. Αλλά οτιδήποτε αφορά την δίωξη κλπ. αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών και των ε, νομότυπων ε, διοκτικών αρχών. Εκεί ακολουθούμε μια προτεραιότητα. Εάν δηλαδή ένα σκάφος συλλάβει πειρατές, τότε εκείνη και το κράτος σημαίας είναι που θα, θα κρίνει αν θα υπάρξει βίωση. Παράδειγμα, απλό, αν πάρω με τη χώρα τη δική μου, αν ένα σκάφος με ολλανδική σημαία πέσει θύμα πειρατείας και ε, διασωθεί από Ολλανδικό σκάφος, τότε η δίωξη θα γίνει στην, στην Ολλανδία. Αρκετοί πειρατές έχουν διωχθεί σε διάφορα κράτη-μέλη. Είχαμε και πιο δύσκολα περιστατικά όμως, όταν είναι άλλες οι σημαίες ευκαιρίας. Το κράτος σημαίας είναι ε, αυτό που παίζει ρόλο, είναι σημαντικό για το σκάφος. Υπάρχει αυτή η σχέση τυπικά. Αλλά τα κράτη-μέλη και τρίτες χώρες που των οποίων πληρώματα συμμετέχουν στην δράση της πειρατείας, που ενέχονται, πολλές φορές θέλουν εκείνα να ε, ασκήσουν τη δίωξη. Καμιά φορά δεν θέλει κανείς να ασκήσει τη δίωξη. Τότε πρέπει να απελευθερωθούν οι πειρατές. Εκεί ε, το κόστος και το ρίσκο, το ρίσκο αυξάνονται για τους επικεφαλείς των πειρατών. Ε, όπως σας είπα ε, στην εντολή μας ε, περιλαμβάνεται και η παρακολούθηση της αλίας παράνομη αλία, το κάνουμε αυτό τώρα για τα μη επανδρομένα σκάφη έχουμε ένα σκάφος το οποίο έχει πάνω τέτοια μη επανδρομένα σκάφη μπορεί να χρησιμοποιηθούν αλλά πιο σημαντικές είναι οι δορυφορικές εικόνες που παίρνουμε και τα αναγνωριστικά ε, αεροσκάφη. Ε, αλλά σίγουρα ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα μη επανδρομένα σκάφη. Ο κύριος Κώστερς. Ευχαριστώ. μια στιγμή λέει ο Πρόεδρος, μια στιγμή. Γιατί υπάρχει μια ερώτηση ακόμα από την κυρία Βάιλερ. Μια ερώτηση για το FBI. Είναι χρήσιμο, χρειάζεται μετά από τις θετικές σας εμπειρίες είναι χρήσιμο να κάνουμε κάτι ανάλογο στην Ευρώπη. Okay. Uh, because we are... Επειδή υπάρχει χρόνος, έτσι κι αλλιώς θα ρωτούσα αν θέλατε δεύτερο γύρο, αλλά αν έχετε και εσείς μια ερώτηση, κάντε τη τώρα. Ναι, και εγώ θέλω μια διευκρίνηση. Είπατε 140 πειρατές ε, είπατε ότι διώχθηκαν και πόσες οργανώσεις ή τελικά μόνο τους δράστες αυτούς που είναι ακριβώς ε, εμπλεγμένοι άμεσα εκείνη τη στιγμή φυσικά με φυσική παρουσία στην πειρατεία μόνο αυτοί διώκονται ή και κάποιες οργανώσεις τους. Ίσως ο αντιστράτηγος να απαντήσει πρώτα σε αυτές τις δύο ερωτήσεις και μετά ο κύριος Κώστερ. Παρακαλώ. Ναι, για το κατά πόσο χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή οργάνωση αντίστοιχη των ε, Ηνωμένων Πολιτειών, ίσως στο μέλλον να γίνει αυτό δυνατό, αλλά είμαστε ακόμα μακριά. Γιατί οι περισσότερες δράσεις είναι εθνικές. Υπάρχει κυριαρχία. Και χρησιμοποιούμε τις προξενικές αρχές όταν πρόκειται για συνεργασία. Τώρα κατά πόσο διώκουμε, δεν διώκουμε εμείς, έτσι, οι χώρες μέλη ε, και στον Μαυρίκιο και στις Εχέλες ε, γίνονται οι διώξεις. Οι αποδείξεις που έχουμε αφορούν άτομα. Οπότε δεν ε, μπορώ να πω ότι διώκουμε οργανώσεις. Μπορεί να έχουμε μια ιδέα για το ποιες είναι οι οργανώσεις τους αλλά οι διώξει γίνονται σε βάρος αυτών που με φυσική παρουσία ήταν στο σημείο της πειρατείας και παραβίασαν τον νόμο. Γι' αυτούς έχουμε αποδείξεις, οπότε αυτούς διώκουμε. Ωραία, ο κύριος Κώστας τώρα. Ευχαριστώ. Ναι, δεν χρειάζεται να επαναλάβω αυτά που είπε και ο αντιστράτηγος, αλλά όντως οι δράστες δεν έχουν κοινωνικά μεγάλο κύρος ε, πάντα, συνήθως προσπαθούν να το αποκτήσουν με εγκληματικές συμπεριφορές. Δεν είναι και πολύ έξυπνοι. Πριν από μερικές εβδομάδες προσπάθησαν να ανέβουν σε μια ισπανική φρεγάτα. Αλλά ήταν ανόητο γιατί αμέσως αποθήθηκαν. Οι άνθρωποι αυτοί, όπως είπε και ο αντιστράτηγος, θα διωχθούν αυτοί στην Ισπανία. Θα γίνει δίκη εκεί. Τώρα βέβαια συνδυάζεται η πειρατεία με την φτώχεια και δεν υπάρχει μία και ίδια λύση παντού για την πειρατεία. Από πού έρχεται η πειρατεία, που απευθύνεται, ποια είναι η πρόλευσή της κτλ. Ε, αυτές οι ερωτήσεις όντως πρέπει να αποτελούν μέρος ενός γενικότερου πακέτου δραστηριοτήτων για να βρεθούν λύσεις και να σταματήσει η πειρατεία. Αυτό σημαίνει φυσικά ότι πρέπει να στηρίξουμε και την κυβέρνηση στη Σομαλία. Έπειτα έχει να κάνει και με την διασπορά της Σομαλίας και γι' αυτό αναφέρθηκε και στο Μαλί ο αντιστράτηγος γιατί είπαμε ότι πολλές φορές η Λία καταλήγει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πάρα πολλοί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πολλούς Ομαλούς. Κένια. Μαϊρόμπι. Εκεί βρίσκονται 500.000 Σομαλοί. Υπάρχει μια τεράστια δηλαδή κοινότητα της Σομαλίας στη χώρα αυτή. Ρωτήσατε για το, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η δράση νέμεσης της μικτής ερευνητικής ομάδας έχει γετικό ρόλο, γιατί συνήθως επικεφαλής είναι ένα εισαγγελέας. Σε αυτή την περίπτωση μόνο ο Λαδός θα μπορούσε να είναι, γιατί ο Γερμανός δεν έχει δικαιοδοσία στα ανοιχτά της θάλασσα. Ενώ ο Λαδό εισαγγελέα, ναι, για λόγους ιστορικούς, γιατί της Ολλανδίας το ναυτικό έχει πίσω του μεγάλη ιστορία. και με πειρατεία και με πλοία, καραϊβική, την εποχή της Ισπανίας κλπ. κλπ. Μεγάλη ιστορία από πίσω δηλαδή. Το θέμα είναι θέμα δικαιοδοσίας. Και δεν ξέρω κατά πόσο στη δικαιοδοσία που δεν υπάρχει βέβαια ακόμα ο Ευρωπαίος εισαγγελέα, αλλά αν υποθέσουμε ότι υπήρχε δεν ξέρω τι δικαιοδοσία θα είχε. Πάντως με κάθε σεβασμό εξακολουθεί να είναι εθνική αρμοδιότητα. Είναι θέμα εθνικής δικαιοδοσίας και εθνικής νομοθεσίας. Με ρωτήσατε και για το TFTP, τη συμφωνία αυτή, που πρόκειται για το πρόγραμμα ανείχνευσης ε, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας πάντα υπάρχει μια σχέση με την τρομοκρατία. Αν ρωτήσουμε το αντίστοιχο πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών και θέλουμε να ζητήσουμε από εκεί κάτι, πρέπει να αποδείξουμε ότι υπάρχει σχέση με την τρομοκρατία. Και πρέπει να αποδειχτεί και οι Ηνωμένε Πολιτείε επίσης θα το εξετάσουν και θα δουν, να δούνε κατά πόσο έχει βάση ο ισχυρισμός μας για σύνδεση με την τρομοκρατία. Εφόσον υπάρχει κάποιο πειρατή και μπορεί να είναι ύποπτος για σχέση με την Al-Shabaab, τότε σίγουρα θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα αλλά πρέπει να υπάρχει απόδειξη. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα για σοβαρά διασυνοριακά εγκλήματα. Όχι. Αυτό το πρόγραμμα είναι μόνο για την περίπτωση της τρομοκρατίας. Η συμφωνία αυτή, η TFTP, είναι πολύ σοβαρή και πολύ ισχυρή για να την καταχραστούμε χρησιμοποιώντας την στην περίπτωση που δεν έχουμε αποδείξεις για τη σύνδεση με την τρομοκρατία. Νιγερία τώρα. Εκεί στις ακτές τη βλέπουμε. Με έχουν ξαναρωτήσει το ίδιο πράγμα. Βλέπουμε να γίνονται ληστείες, όχι μόνο πειρατεία, αλλά και ληστείες στην ε, θάλασσα. Μόλις έξω από το λιμάνι είναι ένα πλοίο και έρχεται κάποιος, ανεβαίνει απάνω, κλέβει ό,τι μπορεί και φεύγει. Θα λέγαμε ότι πρόκειται για ληστεία στη θάλασσα και όχι για πειρατεία στη θάλασσα. Η πειρατεία σημαίνει ότι απαγάγεις τον κόσμο και ότι αναλαμβάνεις εσύ ε, το σκάφος. Τότε πρόκειται για πειρατεία. Νομίζω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με κάνετε όντω να πω πίσω στο 16ο αιώνα, όταν και εμείς οι Πορτογάλοι ε, πολεμήσαμε τους Ολλανδούς και υπήρχε πυρετία στη Σακότρα για παράδειγμα ε, και στην Ιαμένη. Δεν ξέρω αν θέλετε άλλες διευκρινήσεις, άλλες ερωτήσεις. Όχι. Α, παρακαλώ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, έχω απογοητευτεί λιγάκι, παρόλο που είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτά που μας είπατε, αλλά βλέπετε, εμεί θέλουμε να ασχοληθούμε με το οργανωμένο έγκλημα και τις εγκληματικές οργανώσεις. Θέλουμε να καταλάβουμε καλύτερα τη φύση του οργανωμένου εγκλήματος για να το καταπολεμήσουμε, να το αντιμετωπίσουμε, πάση περιπτώσει. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ επικεντρωθήκαμε στην πειρατεία, πιο συγκεκριμένα στον πειρατή το συγκεκριμένο. Που είπατε τότε. εντάξει, συνήθω είναι κάποιος ευάλωτος, φτωχός, ε, ταλέπορος. Ε, αυτός είναι ο δράστης της ε, πειρατείας, αλλά πίσω από αυτό βρίσκεται συνήθως μια ολόκληρη εγκληματική οργάνωση που βγάζει πάρα πολλά λεφτά από τέτοιες επιχειρήσεις. Για μένα λοιπόν λείπει ένας κρίκος. Ξέρετε πολύ καλά, είπατε πιάσατε 140 πειρατές. Ωραία. Πρόεδρος, νομίζω ότι το έχουμε λύσει αυτό. Συγγνώμη, εμφανίζομαι εδώ ξαφνικά όντως στην επιτροπή αυτή, και, αλλά άμα είναι μέχρι τις 6.30 γιατί να μην χρησιμοποιήσω Αν δεν πρέπει, συγγνώμη, συγγνώμη, εντάξει, συγγνώμη αν παρεκκλίνω από τι διαδικασίε. αλλά η Επιτροπή μα θέλει να εξετάσει το οργανωμένο έγκλημα. Να συζητήσουμε λοιπόν για το οργανωμένο έγκλημα και όχι για αυτού του ταλέπορου πειρατέ. Διευκρίνηση, δεν ξέρω, θέλετε μήπως να απαντήσετε. Παρακαλώ. Κύριε Κώστης. Ναι. η πειρατεία στη θάλασσα οργανώνεται όντως από τη στεριά. Της Σομαλίας, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Περιοχή που βρίσκεται υπό την Αλ-Σαμπάμπ. Δεν υπάρχει αστυνομία, δεν υπάρχει δικαιοδοσία. Οπότε με κάθε σεβασμό η επικεφαλής, οι big boys, ε, δεν θα είναι ποτέ στο σκάφος, είναι στη στεριά και προς το παρόν δεν υπάρχει δυνατότητα να πάμε σε αυτή τη στεριά και να επιβάλλουμε τον νόμο, να του συλλάβουμε, να του αντιμετωπίσουμε τέλος πάντων επί τόπου. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Πρώτον, εμείς ως Ευρωπαϊκή Αστυνομική Αρχή δεν έχουμε δικαιοδοσία εκεί πέρα. Δεν έχουμε εκτελεστικές εξουσίες. Δεν μπορούμε να πάμε σε μια χώρα και να κάνουμε συλλήψεις. Είναι δύσκολο το θέμα αυτό. Αναλύοντας όμως τις πληροφορίες που έχουμε, ανταλλάσσοντας πληροφορίες, μπορεί να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ένας από αυτούς τους big boys βγαίνει από εκεί, από αυτή την ασφαλή για αυτόν ζώνη και τότε μπορούμε να παρέμβουμε. Τότε θα το συλλάβουμε. Αυτό περιμένουμε. Δεν έχουμε εκτελεστικές εξουσίες όπως σας είπα, δεν έχουμε δικαιοδοσία να δράσουμε μέσα στην Σομαλία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Εσείς κύριε Τιστράτη έχετε κάτι να προσθέσετε. Νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο ερώτημα, γιατί σχετίζεται με το πώς επιλύουμε το πρόβλημα. Και δεν θα έπρεπε να πολεμούμε μόνο τους πειρατές ε, στη θάλασσα. Είναι να συλλαμβάνουμε μόνο ε, τους ε, μικρούς διακινητές εμπορών και να αφήνουμε τους βαρύνους ελεύθερους. Έτσι λοιπόν, ε, αν θέλουμε να δούμε την πειρατεία σε οργανωμένο έγκλημα, πρέπει να δούμε ποιες είναι οι αιτίε που εξωθούν τους ανθρώπους στην πειρατεία. Και δεν είναι μόνο η ηγεσία. Έχουμε και κόστος όφελος για τους αρχηγούς, αλλά και για τα άτομα. Κάνουν την επιλογή να προβούν σε εγκληματικέ πράξεις. Ξέρουν ότι είναι παράνομο κάτι τέτοιο. Και επειδή δεν υπάρχει και επιβολή του νόμου στη Σομαλία. Δεν υπάρχει ασφάλεια γενικότερα. Δεν υπάρχει καλή διακυβέρνηση γενικά. Ναι, υπάρχει φτώχεια λόγω όλων αυτών, γιατί αν δεν υπάρχει καλή διακυβέρνηση θα υπάρχει και φτώχεια. Πρόκειται λοιπόν αυτό το σύνολο παραγόντων και το βλέπουμε όλο αυτό. Προσπαθούμε να δούμε ποια είναι η αιτία τη πειρατεία και προσπαθούμε ω Ευρωπαϊκή Ένωση να τα λύσουμε όλα αυτά συντονισμένα. Αυτό προσπάθησα να εξηγήσω. Και εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο ρόλο. Εγώ βέβαια στρατιωτικός ε, δεν έχω τη δικαιοδοσία να πάω και να συλλάβω τους ανθρώπους της εξαιρέσεις. Εξήγησα τι μπορώ να κάνω, αλλά υποστηρίζουμε την επιβολή του νόμου. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ευρύτερος οργανισμός, Συμβούλιο Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και Κομισιόν από κοινού κάθονται γύρω από το τραπέζι, εξετάζουν ε, όλε αυτέ τι διαφορετικέ αιτίε και πώ θα τι επιλύσουμε. Νομίζω ότι κάναμε ένα μεγάλο βήμα προ τα μπρο ε, στο να ομοδοποιήσουμε όλα αυτά τα διαφορετικά μέσα. Αλλά μία ακόμη πτυχή που πρέπει να επιδιώξουμε είναι να βρούμε τους αρχηγούς των σημεριών, αυτούς που συνεχίζουν να επενδύουν χρήματα και πληρώνουν ε, αυτούς τους ανθρώπους που μπαίνουν στα σκάφη και κάνουν αυτές τις πράξεις πειρατείας. Δεν έχουμε λύση για αυτό το τμήμα, αλλά τουλάχιστον προσπαθούμε. Αναπτύσσουμε περαιτέρω, γιατί αν πετύχουμε αυτό το συντονισμό μεταξύ ΜΟΝ και Europol και μπορούμε να έχουμε αυτές τις ε, πληροφορίες που θα είναι κατάλληλες για να εντοπίσουμε τους αρχηγούς, τότε θα μπούμε και στις αιτίε. Εν τω μεταξύ προσπαθούμε να βρούμε λύσεις για το ότι δεν υπάρχει επιβολική δικαίου και ασφάλεια. Γιατί εδώ ε, αυτό που προσπαθούν να κάνουν και η αποστολή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άμυνας ε, και Ασφάλειας, ε, αλλά και η ανθρωπιστική βοήθεια. Μάλιστα. Άλλα σημεία, στα διάφορα έχουμε κάτι, αν όχι. Θα συνεδριάσουμε την μόνη φορά, εδώ στις 18 Μαρτίου, από τις 3 ως τις 6.30 το απόγευμα και 19 Μαρτίου από τις 9 το πρωί μέχρι το μεσημέρι και το απόγευμα σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ τους δύο μιλητές για την παρουσία τους και όλους όσους περιβρεθήκατε σε αυτήν την ακρόαση. Καλό βράδυ σε όλους. Thank you